Diamo Καλώς ήρθατε όλοι. Ξεκινάμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Πρώτα-πρώτα μια μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Εάν συμφωνείτε, θα έλεγα να δούμε τα σημεία 6 και 7 πριν από το 5. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, τον κύριο Μογγέλ, και για τον προπολογισμό μετά το 2013. Ο κύριος Μέγγελ θα παραστεί και στην συζήτηση για την κοινή γεωργική πολιτική και εάν ε, μπορείτε να συμφωνήσετε θα δεχτούμε αυτή την αλλαγή στην ημίσια διάταξη. Τώρα, έγκριση των πρακτικών στις 25, της συνεδρίασης 25 και 26 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου του 2011. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις πριν από το τέλος της συνεδρίασης και τα πρακτικά της συνεδρίασης θεωρούνται εγκεκριμένα. Στην ε, σημερινή συνεδρίαση θα έχουμε web streaming. Και επιπλέον σα ενημερώνω ότι ο, ο Επίτροπος, ο κύριος Τσόλο, υπεύθυνο για την Γεωργία για την ανάπτυξη της υπαίθρου, θα παραστεί στην Επιτροπή μας στι 15 Μαρτίου για να παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών, το νομοθετικό πρόγραμμα εργασιών για το 2012. Εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Τσόλος για να μας παρουσιάσει, όπως είπα, το πρόγραμμα εργασιών της Εκτελεστικής Επιτροπής για το 2012. Επιπλέον θα έρθει και ο Επίτροπος ε, Νταλή, Νταλή για την, ε, υπεύθυνο για την υγεία και τη ζωική υγεία στις 12 Απριλίου. Ας σημειώσουμε λοιπόν αυτές τις δύο σημαντικές ημερομηνίε ε, στην ατζέντα μας στις 15 Μαρτίου ο κ. Τσόλος και στις 12 ο κ. Νταλή. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Όλοι έχετε λάβει τον κατάλογο των ψηφοφοριών η Ευρώπη, πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο, ένα νέο πλαίσιο πολιτική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Εισηγητή, ο αντιπρόεδρο Λούτσιαν Νικουλέσκου. Επέφθηνε επί τη ουσία η Επιτροπή Μεταφορών και για την ώρα έχουν υποβληθεί 35 τροπολογίες ε, για την γνωμοδότηση αυτή. Ο εισηγητής έχει ζητήσει να πάρει για λίγο το λόγο θα δώσω λοιπόν το λόγο στον συγκεκριμένο, στον τον κύριο Νικουλέσκου και αμέσως μετά θα ψηφίσουμε. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Θεωρώ ότι όλες ήταν πολύ χρήσιμες και εύστοχες και για αυτό το λόγο θα έλεγα οι συνάδελφοι να τις υπερψηφίσουν. Νομίζω ότι συνολικά θα έχουμε μια καλή έκθεση ποιότητας και ελπίζω ότι η υπεύθυνη Επιτροπή επί της ουσίας, η Επιτροπή Μεταφορών, θα λάβει υπόψη τη δική μας την ε, τοποθέτηση. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο κ. Νικουλέσκου. Και τώρα, αν είστε έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Έτοιμοι. Έχετε τις κάρτες σας. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε. Ένα. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 1. Έναρξη. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Πρόεδρε, θα έπρεπε να αναβληθεί η ψηφοφορία, διότι δεν έχει αρκετό σοσιαλιστέ στην αίθουσα και δυσκολεύτηκε πολύ αυτή η τροπολογία. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία παριθμών 2. 2. Ένα έναρξη ψηφοφορία, Νταντέν. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Ε, συγγνώμη, πέντε. Πέντε. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έξι. Έξι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την υπαριθμόν 7. Έναρξη ψηφοφορία για την 7. Γκουτιέρε Γκαρσία. 7. Πέρα. Εγκρίνεται. 9. Νεντελτσέβα. Έναρξη ψηφοφορία για την υπαριθμόν 9. Έναρξη. Πέρα. Εγκρίνεται. 10. Ντάντζιλα. Έναρξη για την 10. Πέρα, Η παριθμόν 10 εγκρίνεται. 11. Πόλσεν και λοιπή. Άρχεται η ψηφοφορία για την 11. Πέρα. Εγκρίνεται. 12. Έναρξη ψηφοφορίας για την 12. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Έναρξη ψηφοφορίας για την 13. Πέρας. Εγκρίνεται η 13. 14. Ψηφίζουμε την 14. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 15. Έναρξη ψηφοφορία για την 15. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Έναρξη ψηφοφορία για την 16. Πέρας. Εγκρίνεται. Έναρξη ψηφοφορία για την 17. Σκοτά και λυπή. Έναρξη ψηφοφορία για την 17. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία παριθμών 18. 18. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19. Άρχεται η ψηφοφορία για την υπαριθμό 19. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 20. Άρχεται η ψηφοφορία για την 20. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 21. Πέρας. Απορρίπτεται. 22. 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Άρχεται η ψηφοφορία για την 23. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. 24. Πέρας, εγκρίνεται. 25. Άρχεται η ψηφοφορία για την 25. Πέρας. Εγκρίνεται. 26. Άρχεται η ψηφοφορία για την 26. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. 27. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. 28. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Σε δύο τμήματα. Τροπολογία 29 πρώτο τμήμα, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. 29, πρώτο τμήμα, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 29, δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. 30. Τροπολογία υπεριθμών 30. Άρχεται η ψηφοφορία για την 30. Πέρα. Εγκρίνεται. 31. Τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. 32. Άρχεται η ψηφοφορία για την 32. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 33. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Όχι, εκδοτή 35. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία περιθμών 35. Πέρας. Και τώρα, συνάδελφοι, ψηφίζουμε για το τελικό κείμενο ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία, η τελική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον Αντιπρόεδρο Νικουλέσκου. Ωραία. Συνεχίζουμε. Αμέσως περνάμε στο σημείο 6. Ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης. Καλωσορίζω τον Διευθυντή Χόλγκερντ, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη, που θα μα παρουσιάσει πληροφορίε σχετικά με την κατάσταση τη αγορά τη ζάχαρη, που αυτή τη στιγμή γνωρίζει σοβαρή έλλειψη ισορροπία. Θα ξέρετε ότι οι τιμέ ξεπήρασαν τα 1000 δολάρια τον τόνο. Όπω επίση θα γνωρίζετε, η Διαχειριστική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την κοινή οργάνωση αγορά αποφάσισε την περασμένη Πέμπτη βάση πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Εκτελεστικής Επιτροπής να ε, σταματήσει, να πάυσει την ε, επιπλέον καταβολή 500 ευρώ ανά τόνο και να ε, καθορίσει στο μηδέν την ανώτερη ποσότητα των 500.000 τόνων ζάχαρης εκτός ποσόστοσης και σε 26.000 ε, τόνους την ισογλυκόζη. Καθώς και να επιτρέψει εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα σύστημα διαγωνισμού. Κύριε Χέλγκαρτ, θα σας δώσω το λόγο για να μας δώσετε τις πληροφορίες σας και μετά σε όλους τους συναδέλφους θα έχουν να σας κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Κύριε Χέλγκαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. επειδή οι τιμές έχουν είναι πάρα πολύ υψηλέ, οι διεθνεί τιμέ, Είδαμε, διαπιστώσαμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ζάχαρη υφίσταται μια πολύ σοβαρότερη κρίση από ότι η παγκόσμια κρίση ε, ιδιαίτερα επειδή πολλές χώρες από τις οποίες εισάγεται η ζάχαρη ήταν χώρες ε, οι οποίες ε, υπέφεραν από πολέμους και σοβαρά προβλήματα. Τώρα όμως αυτό δεν ισχύει πλέον όσο ισχύει στο πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε δει μία μείωση της ε, τιμής ε, στην αγορά ως αποτέλεσμα της μείωσης της τιμής αναφοράς της ζάχαρης. Έτσι λοιπόν έπεσαν λίγο οι τιμές και πριν από ένα χρόνο καταλήξαμε στα 479 ευρώ ανά ε, η τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις προφορίες που λαμβάνουμε από τον τομέα. Έχει εντωμεταξύ πάλι αυξηθεί η τιμή από αυτή που ανέφερα και οι προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές. Υπό τις συνθήκες αυτές η Κομισιόν έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις, ε, την ικανοποιητική προμήθεια της ευρωπαϊκής αγοράς με ζάχαρη σύστημα είχε μία συγκεκριμένη ποσόστοση για τους λεγόμενους ε, επεξεργαστές πλήρους απασχόλησης, full-time refiners, ε, οι οποίοι ε, ως πρώτη ύλη δεν χρησιμοποιούνταν τα ζαχαρότευτλα, αλλά το, τα, τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου την οποία εισήγαγαν από τρίτες χώρες και την επεξεργασία την έκαναν ε, σε, ε, ε, χωρίς διακοπή. Η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι τόσο ελκυστική λοιπόν με την τρέχουσα τιμή που έχουμε σήμερα σε σχέση με την τιμή της διεθνούς αγοράς, της παγκόσμιας αγοράς. Και επίσης προβλέψαμε ότι θα υπήρχε μία έλλειψη ε, της ποσότητας ζάχαρης, ιδίως αυτής που προέρχεται από τις χώρες ε, ΑΚΕ. Αυτή τη στιγμή το έλλειμμα υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο τόνου ζάχαρης ε, στο τέλος της ε, τρέχουσας εκστρατείας η οποία τελειώνει τον Οκτώβριο τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Έχουμε ήδη αναστείλει την, το δασμό για ζάχαρη προέλευσης από τη Βραζιλία. Αυτό έγινε, η αναστολή του δασμού έγινε ε, τον Αύγουστο, τον περασμένο Αύγουστο, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις εξαγωγές ζάχαρης εκτός ποσοστώσεων και ταυτόχρονα ε, αναστήλαμε όπως σας είπα τους διαδασμούς από διάφορες χώρες εισαγωγής ε, δεδομένου ότι οι εισαγωγές δεν ήταν ε, τόσες όσες χρειάζονταν για να μην σημειωθεί το έλλειμμα, δηλαδή υπήρχε χαμηλός βαθμός εισαγωγών, αναγκαστήκαμε να συμπληρώσουμε ε, την αγορά ζάχαρης για να μην υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα με εγχώρια ευρωπαϊκή παραγωγή 500.000 ε, τόνων ζάχαρης έχοντας ήδη όμως κάνει εξαγωγές 650.000 τόνων ζάχαρης. Έτσι λοιπόν, από ζάχαρη που δεν εμπίπτει στην ποσόστοση, μετατρέπουμε σε ζάχαρη που εμπίπτει στην ποσόστοση και ε, αναστήλαμε και πάλι τους δασμούς ε, ε, σε μηδέν, σε μηδέν, μηδέν ποσοστό έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και πάλι τις εισαγωγές από τρίτες χώρες για να διευκολύνουμε τις εισαγωγές από από, τα, από ζαχαροκάλαμο και δεδομένου ότι οι χώρες που παράγουν αυτή τη ζάχαρη συνήθως πλήρωναν υψηλό δασμό αποφασίσαμε να εξαλείψουμε το δασμό και να εφαρμόσουμε μηδέν ποσοστό δασμού για να διευκολύσουμε αυτές τις εισαγωγές. Θα μου πείτε γιατί δεν διπλασιάσετε το ποσό των 500.000 για να φτάσουμε στο ποσό του ελλείμματος 1 εκατομμύριο. Το θέμα είναι ότι ε, γνωρίζοντας την εμπορία του παρελθόντος θα επιτρέψουμε καταρχάς αυτές τις εισαγωγέ για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αγορά και τι θα χρειαστεί να κάνουμε σε δεύτερο βήμα. Η αγορά της ζάχαρης λοιπόν είναι υποπίεση, ε, έχουμε ένα έλλειμμα, δεν μπορούμε να καλύψουμε απολύτως τις ανάγκες, οι καταναλωτές χρειάζονται ζάχαρη και έτσι μετατρέπουμε ζάχαρη υποποσόστοση σε ζάχαρη εκτός ποσόστοσης για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις εισαγωγές ε, της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο από τη Βραζιλία που είναι ο μεγαλύτερος ε, παραγωγός αυτού του τύπου ζάχαρης και οι δασμοί είναι μηδενικοί. Ευχαριστούμε τον ε, Διευθυντή Ολγκάρτ με τους ομιλητές που έχουν γραφεί ο κύριος Μόρντεϊ. Η κυρία ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τι μπορεί να μας δείξει καλύτερα την παγκοσμιοποίηση. Βλέπουμε τις παγκόσμιες ανταλλαγές προϊόντων διατροφής. Νομίζω ότι η κατάσταση στην Ουγγαρία είναι εύγλωτη η ε, κατάσταση είναι ιδιαίτερη στην Ουγγαρία. Το ίδιο βέβαια βιώνουν και άλλε χώρε. Σήμερα ο Ούγγρο καταναλωτή, ξέρετε, πληρώνει πολύ ψηλέ τιμέ για τη ζάχαρη. Ενώ στην Ουγγαρία είχαμε 800 εργοστάσια παραγωγή ζάχαρη. Αλλά με την ε, ιδιωτικοποίηση και με την παγκοσμιοποίηση των αγορών μείναμε με ένα εργοστάσιο. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πλήρη αυτάρκεια. Αυτό είναι όμως πλέον στο παρελθόν αλλά ας δούμε το παρόν και το μέλλον. Σε καμία περίπτωση οι Ούγγροι δεν θα εγκαταλείψουμε βέβαια την ιδέα ενδεχομένως ε, να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το δικαίωμά μας στην αυτάρκεια, αλλά έχουμε την συγκεκριμένη πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε και αφού πλέον έχουμε ανάγκη και από εισαγωγές, νομίζω ότι θα έπρεπε να μην είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η ζάχαρη ως καύσιμο διότι αυτό συμβάλλει στην άνοδο της τιμής της ζάχαρης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή το γεγονός ότι ένα προϊόν διατροφής χρησιμοποιείται ως καύσιμο. Και βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε ότι και σε κάποιες ε, μικρού μεγέθους οικογενειακές ε, εκμεταλλεύσεις ίσως θα μπορούσε να ισχύσει αυτό, να γίνεται δηλαδή χρήση της ζάχαρης ως ε, καυσίμου, αλλά όχι στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ποια είναι η πρότασή μας. Ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έπρεπε χρήση αυτή να απαγορευτεί. Αυτή είναι η πρότασή μας, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, εμείς θέλουμε να ξαναισχύσει το δικαίωμά μας στη διατροφική επάρκεια και αυτάρκεια, όπως και προείπα. και υπάρχουν και κάποια παγκόσμια ε, συστήματα εμβολιασμού και ανταλλαγή ε, τροφίμων. Ε, θα μπορούσαν κάποιε χώρε να έχουν δυνατότητα να εξέλθουν από αυτά τα συστήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μορβέη, ο κύριο Στέντι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν έχω πια συμφέρον στη, ζάχαρη. Ήμουν παραγωγός ζάχαρης μέχρι την εποχή της μεταρρύθμισης Είχαμε τότε υπογράψει μία συμφωνία στη δεκαετία του 70 στην δέωση της οποίας είχα συμμετάσχει και εγώ. Τώρα πια δεν έχω κανένα προσωπικό συμφέρον. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με την ιδέα των 500.000 τόνων. Καταρχάς, ε, είναι, είναι αυτή η ποσόστοση της εθανόλης ή η ποσόστοση για ε, προϊόντα εκτός τροφίμων. Εμεί πιστεύουμε στον Ηνωμένο Βασίλειο ότι έπαιξε ρόλο και ο καιρός, οι καιρικέ συνθήκες για την κατάσταση της αγορά, τη ζάχαρη. Όσον αφορά τώρα το δασμό, μιλήσατε για 500 ευρώ ανατόνο και εν συνεχεία είπατε 300.000 τόνοι, οι οποίοι θα έρθουν ε, duty free, άνευ δηλαδή, από χώρες είπατε χώρες ΑΚΕ, είπατε τη Βραζιλία, από, από την παγκόσμια αγορά. Εντάξει. Στην ε, Επιτροπή Εμπορικών Συναλλαγών το πράσινο λόμπι είναι πολύ, ε, παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την εξέλιξη των αγορών στη, στη Βραζιλία και ε, Είμαι απογοητευμένο που η μεγαλύτερη ποσότητα θα προέλθει από τη, από τη Βραζιλία και όχι από χώρες ΑΚΕ. Ε, κρίμα. Ε, εγώ μιλάω τώρα ως παραγωγός, ως ε, αγρότης. Η αγορά αποφασίζει πού θα διοχετευθούν τα προϊόντα. Εάν αρχίσουμε εμείς τώρα να περιμένουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε στον κόσμο, να υποδείξουμε στον κόσμο ότι δεν θα πρέπει να καλλιεργούν αυτού του είδους τα, φυτά για παραγωγή ενέργειας, θα διαστρεβλώσουμε την αγορά ενδέχεται εμείς η παραγωγή να προτιμούμε να καλλιεργούμε για παραγωγή ενέργειας τα κατάλληλα, τις ε, κατάλληλες καλλιέργειες. Εμείς δεν είμαστε φιλανθρωπικό, φιλανθρωπικές κοινωνίες, πρέπει και να επιζήσουμε. Το κάνουμε για τα εισοδήματά μας. Άρα λοιπόν λοιπόν εμείς έχουμε καλλιεργήσει ε, ε, φυτά, ε, χρόνια για την παραγωγή ενέργειας, για την αντικατάσταση του πετρελαίου κλπ. κλπ. Λοιπόν δεν είναι δυνατόν να μας υποδείξει η Κομισιόν τι θα καλλιεργήσουν και ποιοι, διότι αυτό εναπόκειται στις αγορές. Οι αγορές υποδεικνύουν, οι αγορές οδηγούν τι θα καλλιεργήσουμε και πού θα διοχετευτούν. Η τιμή της ζάχαρης ε, ανέβηκε ε, σημαντικότατα, το είδαμε και στην ε, Ρωσία, την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάρκια Παρ' όλα αυτά ανεβήκαν οι τιμές ηλικιωδώς. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Κομισιόν δεν πρέπει να παρέμβει στο να καθοδηγεί την αγορά. Ευχαριστώ, ο κύριος ε, Γκλάτεμφελτ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Με βάση τα πρόσφατα γεγονότα, πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που δεν εγκρίναμε τη μεταρρύθμιση της ζάχαρης. Γιατί τα πρόσφατα γεγονότα και η μεταρρύθμιση της ζάχαρης έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους, ε, πρόδειλη σχέση. Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση της ζάχαρης ε, δεν ευωδόθηκε, δεν ολοκληρώθηκε, αλλά μας δείχνει σήμερα η κατάσταση για ποιο λόγο είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αυτάρκης σε ό,τι αφορά τα σημαντικότερα τρόφιμα, τα σημαντικότερα προϊόντα διατροφής. Ελπίζω να μην ε, αφαιθεί κατά μέρο αυτό το θέμα και όταν ε, μάλιστα ψηφίσουμε για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ο φίλος ε, Άλμπερτ Ντες είναι αυτός ο οποίος έχει συντάξει τη σχετική έκθεση την οποία και θα ψηφίσουμε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις προς την Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια αμφιβολία που έχω. Φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης που είναι κατεστημένες σε αρκετέ χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίε συμπεριφέρονται κατά τρόπο που κανείς θα μπορούσε να θεωρεί συμπεριφορά καρτέλ. Κάποιες φορές ε, βλέπουμε διπλάσια τιμή πώληση τη ζάχαρη σε σχέση με άλλε χώρες μέλη της Ένωσης και μάλιστα σε κάποιες χώρες της Ένωσης αυξήθηκε σημαντικά η τιμή της ζάχαρης όταν μετά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης έκλεισαν εργοστάσια στις χώρες αυτές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως αποστολή να εκπροσωπεί και τα συμφέροντα των καταναλωτών, όχι μόνο να εγγυάται τον ανταγωνισμό. Θέλω, θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτή την κατάσταση καρτέλ. Είναι απαράδεκτο σε κάποιες χώρες η τιμή της ζάχαρης να είναι διπλάσια παρότι προέρχεται από τα ίδια εργοστάσια με τα οποία τροφοδοτούνται και, από τα οποία τροφοδοτούνται και άλλες χώρες. Σε ό,τι αφορά τώρα την ισογλυκόζη νομίζω ότι οι ποσοστώσεις πρέπει να αυξηθούν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστική παραγωγή ισογλυκόζης ως ευρωπαϊκού προϊόντος από τον αραβόσιτο ε, παραδείγματος χάρη. Σε πολλές περιοχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν καλλιέργειες αραβοσίτου και τα εργαστάσια μεταποίησης χρειάζονται χαμηλής ε, τιμής ισογλυκόζη. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε. Θα πρέπει να το σκεφτούμε γιατί Είμαστε στην ε, περιοχή πριν τη φύτευση, ε, του, στην ε, φάση πριν τη φύτευση του αραβοσίτου και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προσπίσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρίτη παρατήρηση τώρα, ή μάλλον ερώτηση, αν μου επιτρέπετε σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις των εργοστασίων εξευγενισμού της ζάχαρης, ραφιναρίσματος. αυτά τα εργοστάσια τα οποία λαμβάνουν μεγαλύτερες ποσοστώσεις είναι αυτά που μπορούν να ε, εξευγενήσουν τη ζάχαρη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Μιλάμε για κάποιες μεταποιητικές βιομηχανίες από ζαχαρότερα και νομίζω ότι αυτές μπορούν να εγγυηθούν στις χαμηλότερες τιμές. Ο κύριος Λάιον, George uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ορισμένες ερωτήσεις προς τον κύριο Χόλγκαρτ για να ε, καταλάβω ακριβώ ε, το υπόβαθρο αυτού του προβλήματος. Ε, ανέφερε ότι έχουμε ένα έλλειμμα στην ευρωπαϊκή αγορά ενός εκατομμυρίου τόνων. Οφείλεται αυτό στην αύξηση της ζήτησης ή στην μείωση της παραγωγής. Ποια είναι τα αίτια. Ε, αναφέρθηκε και το θέμα του καιρού τον, ε, και ότι επειδή το κρύο ήταν ε, πολύ έντονο στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε η παραγωγή κατά πολλούς χιλιάδες τόνους ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αυτό είναι μία ακραία περίπτωση, μία μοναδική περίπτωση ή είναι ένα σενάριο το οποίο επαναλαμβάνεται, δηλαδή ε, σημειώθηκαν λάθη στο παρελθόν και τώρα δεν, να, να δεν υπάρχει επάρκεια ζάχαρη στην ευρωπαϊκή αγορά. Ε, εάν είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει επαναληφθεί, θα πρέπει να το εξετάσουμε εμπεριστατωμένα και θα πρέπει να καταλάβει και η δική μας Επιτροπή ε, σαφώς στα αίτια αυτού του προβλήματος. Grazie George. E adesso l'onorevole Ο κύριος Ρούμπιξ. Μετά ο κύριος Νταντέν και μετά η Νιώ. Έχω. Ευχαριστώ. Η κατάσταση έχει ως εξής. Εμείς τώρα έχουμε διαβάσει την Επιτροπή από το Συμβούλιο, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο λέει σαφέστατα ότι η μεταρρύθμιση της ζάχαρης απέτυχε. Και οι ψηφοφόροι στη Λετωνία ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έκλεισαν τα εργοστάσια ζάχαρης απολύθηκαν εργαζόμενοι και παραγωγοί οι οποίοι καλλιεργούσαν ζαχαρότευτλα δεν συνέχισαν αυτήν την διαδικασία. Κάθε φορά που αντιμετωπίζω ψηφοφόρους με ρωτούν λοιπόν γιατί σημειώθηκαν αυτά τα γεγονότα, αυτή η κακή εξέλιξη. Ήθελε λοιπόν να σας ρωτήσω εάν αυτή η κατάσταση της, ε, ε, του, του, του, του ραφιναρίσματος της ζάχαρης σταμάτησε μετά από πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επειδή το αποφάσισαν οι χώρες μεμονωμένα. Ρωτώ λοιπόν και πάλι, σταμάτησε η παραγωγή λευκής ζάχαρης, της ραφιναρισμένης ζάχαρης λόγω πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλήξαμε σε αυτή την παταγώδη αποτυχία και αρνητική κατάσταση. Πολλοί παραγωγοί έχουν μεταξύ εκφράσει την επιθυμία τους να ξεκινήσουν και πάλι την παραγωγή ζάχαρης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εξ ονόματός τους, εξ τους, θα υπάρχουν ποσοστώσεις μετά το 2013 ή όχι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρία ερωτήματα θέλω να θέσω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να μας πει ποιος είναι ο όγκος της ε, ζάχαρης που παράγεται, μάλλον που παραγόταν στην Ευρώπη το 2005 και το 2010. Όγκος εισαγόμενος 2005 και όγκος εισαγόμενος 2010 και αν η ανάλυση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την εξέλιξη με βάση αυτά που μας είπε το 2006, εάν αυτό αποδίδει, οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα του τομέα της ζάχαρης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μία ερώτηση προς την κυρία Μόρβε από την Ουγγαρία. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι είπε από ό,τι κατάλαβα, είπατε ότι έχετε Α, ναι, δεν κατάλαβα καλά. Οχτώ δηληστήρια έχετε, δηλαδή στάση επεξεργασία ζάχαρης, όχι 800. Ε, λοιπόν, Ας μην ξεχνάμε ότι τα ζαχαρότευτλα έχουν θαυμάσια απόδοση και δεν θα πρέπει να τα πετάμε ε, σε χωματερές όταν έχουμε μία πλεονάζουσα παραγωγή ζαχαροτεύτλων. Είναι ένα θαυμάσιο προϊόν, καλλιεργήσιμο προϊόν και πρέπει τα εργοστάσια ε, παραγωγής και επεξεργασία ζάχαρης να βρίσκονται κοντά στις τοποθεσίες εκείνες όπου καλλιεργούνται ζαχαρότευτλα. Grazie onorevole Agnon. E adesso a chiudere gli interventi l'onorevole Ia. A te. Poi daremo la parola alla Commissione. Και μετά θα έχουμε πάλι το Γενικό Διευθυντή. Ευχαριστώ. Μία συμπληρωματική ερώτηση. Γιατί ε, θα θέλαμε να ξέρουμε πώς εκτιμά τις τιμές στην παγκόσμια αγορά η Κομισιόν. Δηλαδή πώς κάνει την εκτίμηση με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα ή ε, κάνει τις εκτιμήσεις της ε, έτσι ώστε να μπορέσει να προβλέψει και μακροπρόθεσμα της ε, εξελίξεις των τιμών της ζάχαρης. Θα πρέπει να αποφασίσουμε την δομή της αγοράς ζάχαρης τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ ανήκω σε αυτούς που λένε ότι όταν υπάρχει μια παγκόσμια αγορά για αγροτικά ε, προϊόντα, το καλύτερο που μπορούμε να επιτύχουμε είναι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από την Κομισιόν πώς πιστεύω θα εξελιχθεί στο μέλλον η αγορά και πώς κάνει αυτές τις εκτιμήσεις. Ο, ο κύριος Μποβέ. Euh, Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο μετά από τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δομή, για τη δομή η διάρθρωση αν θέλετε των παραγωγών ζάχαρης ανά τον κόσμο. Μετά από αυτά που είπε ο Μισελ Νταντά, ε, την ερώτηση που έκανε για τον όγκο, νομίζω ότι καλό θα ήταν και ενδιαφέρον να μας δώσει η Επιτροπή λίγο ε, το τοπίο, δηλαδή ποιοι παράγουν ζάχαρη. Ευρώπη, Βραζιλία και Βραζιλία. Δηλαδή, ε, είναι σημαντικό να έχουμε κάποια δεδομένα πάνω σε αυτά γιατί σήμερα δεν μιλάμε για αγορές από χώρα σε χώρα, αλλά μιλάμε για αγορές πολυεθνικών που κυρίως βρίσκονται στη Βραζιλία με ποσότητα παραγωγών στην Ευρώπη. Πριν καν δηλαδή ξεκινήσουμε συζητήσεις στους επόμενους μήνες ίσως ή έστω ε, τα επόμενα χρόνια με τις χώρες Μερικοσούρ αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το έχουμε λύσει με σαφή τρόπο για να μην ξαναβρεθούμε στην κατάσταση, για αυτόν τον τομέα όπως και για άλλους πολλούς, η γεωργία, η παραγωγή ε, ζάχαρης, οι αγρότες ουσιαστικά είναι ένα νόμισμα συναλλάγματος αν θέλετε σε σχέση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Σε ευχαριστώ Ζωζέ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, Διευθυντή, κύριο Χέλγκαρτ. Κύριε Χέλγκαρτ, πολλές ερωτήσεις, ελπίζω να καταφέρετε να απαντήσετε και σύντομα σε όλες αυτές. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους όσους έθεσαν ερωτήσεις που καταδεικνύουν την περιπλοκότητα της αγοράς ζάχαρης. Καταρχάς, ε, να, να σας θυμίσω, γιατί έγινε αυτή η μεταρρύθμιση. Είχαμε, ε, την κάναμε για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είχαμε αποφασίσει ότι από τις 48 πιο φτωχές χώρους ε, του κόσμου θα θέλαμε να ενισχύσουμε τις εισαγωγές και να απαλλαγούμε από το παλιό καθεστώ των χωρών ΑΚΕ, ε, το οποίο λειτουργούσε βάσει συγκεκριμένων ποσοστώσεων και να δώσουμε την ευκαιρία στι φτωχότερε χώρε να αυξήσουν τι εξαγωγέ του προ εμά. Οπότε το 2005-2006 βαθμιαία ε, μηδενίσαμε τους δασμού για τις εξαγωγές από αυτές τις χώρες. Ο δεύτερος λόγο για τον οποίο έγινε αυτή η μεταρρύθμιση τη αγορά και συναφεί προσαρμογέ ήταν επειδή το, η ζάχαρη ποιότητος γάμα πιστεύαμε ότι θα, θα πρέπει να εξάγεται ελεύθερα στην παγκόσμια αγορά μαζί με εξαγωγές 1,3 εκατομμυρίων τόνων ε, που δεν υπόκεινταν σε εξαγωγικούς δασμούς η Αυστραλία ή η Ταϊλάνδη έκαναν μία αγωγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου εναντίον μας και χάσαμε στο πάνελ αυτό διότι είπαν ότι το, η ζάχαρη κατηγορίας Γ, C, θα πρέπει να θεωρείται ως υπό επιδοτούμενη ζάχαρη και δεν μπορούσε να ε, ε, εμπέσει στο καθεστώς της ζάχαρης κατηγοριών Α και Β. Είδαμε λοιπόν αυξημένες εισαγωγές λόγω των αποφάσεων που πήραμε, οι οποίες βασμιαία θα μείωναν τη δικιά μας παραγωγή, θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στις δικές μας παραγωγές και εξαγωγές και ε, εφόσον χάσαμε και στον ΠΟΕ, ε, δώσαμε τη δυνατότητα στον τομέα να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, στο νέο καθεστώ και είχαν τελείω ελεύθερη επιλογή, δηλαδή κάθε εμπορευόμενο, ε, κάθε παραγωγό, συγγνώμη, ε, κάθε βιομηχανία σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε τη δυνατότητα, λαμβάνοντας μία αποζημίωση 2.700 ευρώ τόνο να πάυσει την παραγωγή. Ήταν μια πολύ γενναιόδορη προσφορά. Και γιατί ήταν γενναιόδορη, διότι είδαμε ότι ο βιομηχανικός τομέας, ο τομέας γενικά, δεν ήθελε να συμμετάσχει. Υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις να συμμετάσχουν σε αυτή την επιλογή και από 18 σε 14 εκατομμύρια τόνους έπεσε η ποσότητα υπό ε, ποσοστώσεις, που υφίσταται, που εμπίπτει σε ποσοστώσεις. Αυτοί τώρα που επέλεξαν να τοποθετηθούν εκτός ε, του, της αγοράς ήταν και οι λιγότερο αποδοτικοί. Οι καλύτερες μονάδες, οι καλύτερες βιομηχανίες μπόρεσαν να προσαρμοστούν και να αρθολογήσουν την, την παραγωγή τους με το βέλτιστο τρόπο. Και τώρα έχουμε μια κατάσταση όπου η αγορά λειτουργεί πολύ πιο ανταγωνιστικά και επικεντρώνεται κυρίως σε αυτές τις ε, περιοχές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι πιο συμφέρον το κόστος παραγωγής. Ακούσαμε επίσης, και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, ότι ενδέχεται η Κομισιόν ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποχρέωσε ε, τους παραγωγούς να εφαρμόσουν αυτό το καθεστώς των ποσοστώσεων. Όχι, εμείς τους δώσαμε την επιλογή να συμμετάσχουν ή όχι μέσα στο καθεστώς αυτό. Επειδή λοιπόν είχαμε αυτή τη συμφωνία από την πλευρά των εισαγωγών, δεν μπορέσαμε να αποθεματοποιήσουμε ε, τους αναγκαίους ε, τόνους ζάχαρη για τους ε, επεξεργαστές λευκής ζάχαρης. Είναι γεγονός ότι σήμερα τα ζαχαρότευλα είναι πιο ανταγωνιστικά από τι στο διότι τώρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για τη ζάχαρη ποιότητος Β, η οποία έχει μια μικρά περίοδο σχετικά εμπορίας, αλλά στην υπόλοιπη περίοδο, ε, εκεί όπου δεν χρησιμοποιούν, οι μονάδες που δεν χρησιμοποιούν ζαχαρότευτα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζαχαροκάλαμο, που τους δίνει έναν υψηλότερο βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επεξεργαστές ζάχαρης που με συνεχή λειτουργία μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν μία προσφορά βάση της οποίας τους τρεις πρώτους μήνες της εκστρατείας Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ε, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο μπορούσαν να ζητήσουν πιστοποιητικά προέλευσης για να ξέρουν ακριβώς ε, τις, ε, από πού ε, προήλθε η πρώτη ύλη, αν ήταν ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαμο. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο τομέας είναι πολύ πιο ισχυρός και περιέργως στην, στο παρελθόν είχαμε ποσοστώσεις σε εθνικό επίπεδο και τότε οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών ήταν ελάχιστες ε, κατά κάποιο τρόπο οι αγορά, οι αγορές ε, λειτουργούσαν σε στεγανά το μόνο που απασχολούσε τους, ε, ε, ε, τον τομέα ήταν η ζάχαρη να είναι σε αρκετά χαμηλή τιμή, σε τόσο χαμηλή τιμή ώστε να μην είναι ανταγωνιστικές οι εισαγωγές. Αυτή τη στιγμή έχει, έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές τιμών. Σε κάποιο κράτος μάλιστα είναι διπλή η τιμή της ζάχαρης από, τη ένα άλλο. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Να διορθωθεί. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει καλύτερη ισορροπία Σήμερα στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία ε, υπάρχει πλεόνασμα ζάχαρης και βεβαίως η, η, τιμή είναι χαμηλότερη ενώ ελληματικές χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία ε, όπου δεν υπάρχει επάρκεια ζάχαρης οι τιμές είναι υψηλότερες. Ε, διότι τώρα όμως σε αντιστάθμισμα πρέπει να αντιληφθούμε ότι γίνονται ε, μεγάλες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών ενώ στο παρελθόν σχεδόν δεν γινόντουσαν. Υπάρχει η θεωρητική δυνατότητα στον κανονισμό να μεταφέρουμε ζάχαρη εκτός ποσοστώσεων σε ζάχαρη εντός ποσοστώσεων. Ε, κανένας δεν είναι τόσο τρελός ώστε να πληρώσει 500 ευρώ ανά τόνο για να κάνει αυτή τη μεταφορά. Θεωρητικά, άμα το θέλει κάποιος, έστω και τρελός, μπορεί να το κάνει ε, ο μόνος τρόπος που που έχει οικονομική λογική που μπορεί να γίνει αυτή η μεταφορά από εκτός εντός είναι όταν ο δεσμός είναι μηδέν. Τώρα το ερώτημα από πού θα πάρουμε αυτούς τους 500.000 τόνους ε, και το ερώτημα εάν αυξήθηκε η ζήτηση, μειώθηκε η παραγωγή και σημειώθηκε αυτό το έλλειμμα. Πρέπει να απαντήσω αρνητικά και στις δύο ερωτήσεις. Η ζήτηση στην αγορά, στην ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει αλλάξει είναι στο ίδιο ε, επίπεδο. Η παραγωγή ζάχαρης ε, έχει καλυφθεί, δεν, δεν υπάρχει μείωση. Ε, γιατί λοιπόν υπάρχει το έλλειμμα. Υπάρχει το έλλειμμα επειδή υπάρχουν λιγότερες εισαγωγές από ζάχαρη εκτός ποσοστώσεων. Οι ποσότητες ζάχαρης εκτός ποσοστώσεων είναι πολύ λιγότερες φέτος ε, από ό,τι πέρσι. Ε, πέρσι είχαμε 4,6 εκατομμύρια περίπου τόνους ζάχαρης εκτός ποσοστώσεων. Φέτος έχουμε 3 με 3,5 εκατομμύρια τόνους. 3,2 νομίζω εκατομμύρια τόνους. Αυτή η ζάχαρη εκτός ποσοστώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέσσερις σκοπούς. Πρώτον, ή να εξαχθεί, εάν το επιτρέψουμε, σας είπα, επιτρέψαμε εξαγωγές 650.000 τόνων, ή να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοεθανόλης 1,2 εκατομμύρια τόνοι. Τρίτον, να χρησιμοποιηθεί για τη χημική βιομηχανία για να επιτρέψει στη χημική βιομηχανία να ανταγωνιστεί τους ανταγωνιστές της στην παγκόσμια αγορά και να χρησιμοποιήσει τη ζάχαρη ως πρώτη ύλη με τον ίδιο τρόπο που τη χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές της στην παγκόσμια αγορά. Και η τέταρτη δυνατότητα είναι να μεταφερθεί ως ποσόστοση για την παραγωγή του επομένου έτους. Αυτή η οψιόν για του χρόνου ε, δεν θα έχει καμία επίπτωση για το έλλειμμα που, που σημειώνεται. Γι' αυτό θέλουμε να χρησιμοποιηθεί πλήρως η ποσόστοση. Οπότε αντί να επιτρέψουμε περισσότερες εξαγωγές, 350.000 ε, τόνους, ε, τις ε, τροποποιούμε σε ζάχαρη εντός ποσοστώσεων. Τώρα, στο κείμενο του Συμβουλίου και στο κείμενο του κανονισμού, άρθρο 100, 187, λέει και παραθέτω δημητριακά, ρύζι, ζάχαρη, γάλα και γαλακτομικά ή αναφορές τιμών όταν φτάσουν σε ένα επίπεδο όπου υπάρχει ο κίνδυνος τρέβλωσης της κοινοτικής αγοράς και αν υπάρχουν ε, Υπάρχουν ενδείξει ότι αυτή η διαστρέβλωση, η στρέβλωση της αγοράς θα συνεχιστεί, η Κομισιόν, η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εάν οι τιμές, οι παγκόσμιες τιμές δείχνουν ένα επίπεδο που μπορεί να δημιουργήσει στρέβλωση της αγοράς, η Κομισιόν μπορεί να παρέμβει. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε, αποφασίσαμε να υπάρξει αυτή τη στιγμή ε, ε, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες 300 300.000 τόνους προς το παρόν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μετά να ανεβάσουμε τους 300 τόνους εισαγωγή 300.000 σε 500.000 και βλέπουμε. Έχουμε λοιπόν μία υποχρέωση να καλύψουμε το έλλειμμα της εσωτερικής ε, αγοράς. Ήταν άλλο ερώτημα που μετέθη, αν μπορούμε ή πρέπει να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο αυτάρκειας. Κοιτάξτε, ναι, Συνήθως για προϊόντα όπως είναι το ε, λάδι για παράδειγμα έχουμε κάποια αρκετή παραγωγή αλλά αν ε, αυτό δεν ισχύει για κάποια άλλα τρόφιμα αν δεν έχουμε αυτά και θα εξαρτώμεθα από ε, τις εισαγωγές η φιλοσοφία μας είναι η αγορά είναι, να είναι αυτή η οποία θα καθορίσει κατά πρώτο και κύριο λόγο την παραγωγή για να μπορεί να υπάρχουν εμπορικέ συναλλαγέ και ε, στον τομέα των εξαγωγών και στον τομέα των εισαγωγών. Άρα ουσιαστικά το θέμα είναι το εξή. Πέτυχε δεν πέτυχε η μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση δεν έχει αποτύχει. Εάν δείτε τι κατάσταση είχαμε να αντιμετωπίσουμε το 2005, οπότε θα υπήρχαν λιγότερες δυνατές εξαγωγές και περισσότερες εισαγωγές Άρα τότε, όταν μπορούσαμε πλέον να προβλέψουμε την κατάσταση ότι οι τιμέ τη αγορά θα εξακολουθούσαν να είναι πολύ χαμηλότερε από αυτέ της Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλάβουμε ότι έπρεπε να γίνει μεταρρύθμιση. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω, όχι πριν από πολλά χρόνια, η τιμή στι αγορέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τριπλάσια από το επίπεδο της τιμής παγκόσμια αγορά. Τριπλάσια. Και μετά τη μεταρρύθμιση, διπλάσια. Σήμερα, λόγω των εξελίξεων στην αγορά, η κατάσταση διαφέρει εντελώς η τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ίση ή ίσως και χαμηλότερη από αυτή τη παγκόσμια αγορά. Τώρα το ερώτημα θα συνεχιστεί αυτό. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω μεγαλύτερη σοφία από τους παρισταμένους, το αντίθετο θα έλεγα, άρα δεν μπορώ να σας κάνω μία στέρη εκτίμηση. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι αυτό που βλέπουμε στην παγκόσμια αγορά, είτε στον τομέα των δημητριακών, των ελαιούχων σπόρων, είτε άλλων γεωργικών προϊόντων, αυτό που βλέπουμε είναι σημαντική μεταφορά ε, μεταξύ της ε, ζήτησης και της προσφοράς. Δηλαδή υψηλότερες τιμές ε, στην παγκόσμια αγορά, μακροπρόθεσμα, σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε δει τα τελευταία 20, 30 και περισσότερα χρόνια. Επομένως θα υπάρξει πραγματικά μία σημαντική προσαρμογή τιμών, κατά την άποψή μου. Και θα ε, περιλαμβάνει αυτό και τη ζάχαρη. Γιατί? Γιατί η ζάχαρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Βραζιλία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω γνωρίζουμε, όχι μόνο για την παραγωγή ζάχαρη προ κατανάλωση, αλλά και για παραγωγή βιοεθανόλη. Και αν έχουμε 100 δολάρια τιμή ενέργεια ανά βαρέλι πετρελαίου, αυτό αποτελεί κίνητρο ώστε η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμα να χρησιμοποιηθεί περισσότερο για την παραγωγή βιοθανόλης παρά για την παραγωγή ε, βρώσιμη ζάχαρη. Δεν ε, θέλω να το λάβετε αυτό υπόψη σε ένα σενάριο που θα γίνει οπωσδήποτε, αλλά σα το λέω γιατί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι υψηλότερε τιμέ όχι μόνο για τη ζάχαρη αλλά και για άλλα προϊόντα. Κύριε Πρόεδρε, μακρηγόρησα, μπορεί να ξέχασα, ελπίζω όχι, να απαντήσω και σε ορισμένα ερωτήματα. Αν έχω ξεχάσει θα επανέλθω. Αλλά θέλω να πω, αν ναι, και ένα τελευταίο ερώτημα, εμείς δεν θεωρούμε ότι με μια αύξηση των ποσοστώσεων ισογλυκός μπορεί να ληφθεί υπόψη και να γίνει έτσι ε, απομονωμένα. Ε, σας επανθυμίζω ότι πρόσφατα έγινε μεταρρύθμιση και όπως είπαμε οι ποσοστώσεις ε, λήγουν το 2015. Άρα είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Υπό τις παρούσες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη των αγορών που αλλάζουν, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τις ποσοστώσεις ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στέρη, θέλετε το λόγο, αλλά λίγο σας παρακαλώ, γιατί έχουμε πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υπενθυμίσω στην Κομισιόν ότι όταν προσυπογράψαμε το πρωτόκολλο τη ζάχαρη δεκαετία του 70, οι παγκόσμιε τιμέ αγορά ε, ήταν υψηλότερε από αυτή που προτείναμε εμεί και υπήρξε δέσμευση ε, χωρών ΑΚΕ και χωρών Ευρωπαϊκή Ένωση για να εγγυηθούν την αγορά. Και δεύτερον, δεν είχε επιλογή ο παραγωγός. Εκπλήσουν από αυτό που λέει η Κομισιόν. Και πρέπει να σας πω ότι σίγουρα σε κάποιες ε, χώρες οι μεταμπητές, οι επεξεργαστές είχαν το μονοπόλιο. Αποφάσισαν τι τους συνέφερε περισσότερο. Όχι που καλλιεργούνται τα καλύτερα προϊόντα. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη της Κομισιόν, κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση, φυσικά και το Διευθυντή, κύριο Χέλγκαρτ, αλλά αν μου επιτρέπετε μία μικρή παρατήρηση, κύριε Χέλγκαρτ, μετά τη μεταρρύθμιση του 2005 έχουν κλείσει πάνω από 80 εργοστάσια στην Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα μάθημα για τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε ένα μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα γιατί δεν είναι δυνατό να προκαλείται ένας τόσο δραματικός οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος όπως αυτός που έγινε με τη μεταρρύθμιση στον τομέα της ε, ζάχαρης και προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πληγές μας τώρα. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Θα παρακαλέσω για μια ακόμη φορά τον Διευθυντή κύριο Χέλγκαρτ να μας ενημερώσει για την εφαρμογή του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φρούτα στα σχολεία. Ε, φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις για, για την έναρξη του προγράμματος αυτού. Θέλω να ξέρω λοιπόν αν τα πράγματα βελτιώθηκαν, τι γίνεται σήμερα και τι βελτιώσει θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και για το μέλλον. Κύριο Χέλγκαρτ, για μια ακόμη φορά έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα Φρούτα στα σχολεία. Και Ελπίζω να έχουμε και χρόνο να δούμε και τα άλλα σημεία τη ημερησία διάταξη και δει την έκθεση Albert Dess, Οπότε θα παρακαλέσω και του συναδέλφου για αυτό το θέμα να μην μακρηγορήσουν. Περιμένουμε με μεγάλη υπομονησία την έκθεση Dess. Κύριο Χέλγκαρτ, να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο για τη ζάχαρη. Αυτοί που δεν παράγουν σήμερα ζαχαρότεφλα μπορούν να, παρα... να παράξουν δημητριακά ή ελαιούχου σπόρου και να τα καταφέρουν καλύτερα από ό,τι όταν παρήγαγαν ε, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Οι συγκεκριμένοι αγρότε που άλλαξαν δηλαδή καλλιέργεια τα καταφέρουν καλύτερα σήμερα σε σχέση με το παρελθόν και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το πρόγραμμα για τη διανομή φρούτων στα σχολεία. Αυτό προέκυψε από τη μεταρρύθμιση τη κοινή οργάνωση αγώνα με των οποροκυπευτικών. Υπήρξε έντονη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την ευγνωμονούμε, ευγνωμονούμε το Κοινοβούλιο για τη εισφορά και την υποστήριξη και είχαμε το ποσό των 11 εκατομμυρίων, το είχαμε θέσει κατά μέρο του προβλησμό για το πρόγραμμα αυτό και η κατανομή του ποσού έγινε με βάση τις ανάγκες ε, και τα αιτήματα των κρατών μελών. Κάποια κράτη-μέλη δεν ήθελαν καν να λάβουν μέρος για τον ένα ή τον άλλο λόγο, αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη ήθελαν. Άρα είχαμε 23 συνολικά κράτη-μέλη που ήθελαν να ενταχθούν το 2009 και το 2010 σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, το πλεόνασμα που δεν χρησιμοποιήθηκε από τους μη συμμετέχοντες επαναδιανεμήθηκε στους λοιπούς. Σε αυτούς δηλαδή που ενδιαφέρονταν να διεξαγάγουν αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσό αναδιανεμήθηκε συνεπή αυτού. Τώρα, λόγω των ε, διαφόρων προβλημάτων που υπήρξαν από πλευρά υλικοτεχνική ε, υποδομή, εφαρμογή, κάποια διοικητικά ζητήματα και αιτήσει για συγχρηματοδότηση, απέτηση μάλλον για συγχρηματοδότηση που πρέπει να το υπενθυμίσω, Υπάρχει συγχρηματοδότηση της τάξης του 50% από τα κρατημέλη υποκανονικές συνθήκες για αυτό το πρόγραμμα και χρηματοδότηση 25% στο πλαίσιο των χωρών συνοχής, όπως αποκαλούμε. Άρα ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 90 εκατομμύρια ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή μετά των εθνικών κρατών που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 156 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον εθνικό προπολογισμό. Λόγω αυτού ακριβώ του θέματος, λόγω δηλαδή τη σύγχρηματοδότηση, για να σα το τονίσω αυτό, στη Γερμανία, στα 16 κρατήδια, τα 7 μόνο να έχουν επιλέξει να συμμετέχουν. Λόγω ακριβώ αυτή τη πτυχή, της συγχρηματοδότηση, που ήταν ένα από του λόγου. Μια άλλη πτυχή ήταν κάποια κριτική που ασκήθηκε για το μεγάλο φόρτο εργασία ό,τι αφορά τον έλεγχο, ό,τι αφορά τα διοικητικά και εδώ νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κλασικό πρόβλημα. Από τη μία πλευρά δηλαδή προσπαθούμε να προωθήσουμε έναν καλό στόχο που βρίσκει τους πάντες σύμφωνους, αλλά από την άλλη πλευρά τα χρήματα των φορολογουμένων θέλουμε να χρησιμοποιηθούν με το σωστό τρόπο για να μην υπάρξουν καταχρήσεις και πρωτοσέλιδα εφημερίδες που δεν θα μας άρεσαν καθόλου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανάγκη συνεχούς εξισορρόπησης από τη μια εκπλήρωση του στόχου και αφετέρου τήρησης των απαιτήσεων για την ε, χρηστή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Τι συνέβη το πρώτο έτος, 2009-2010. Δεν δαπανήθηκε το πλήρες ποσό των 90 εκατομμυρίων, γιατί είχαμε αυτές τις καθυστερήσεις και αυτά τα προβλήματα. Μόνο το 37% δαπανήθηκε, δηλαδή 33 εκατομμύρια περίπου λίγο πάνω από το 1 τρίτο, δηλαδή των 90 εκατομμυρίων. Φέτος, 2010-2011, τα πράγματα φαίνονται πολύ πιο λαμπρά, πολύ πιο αισιόδοξα. Μάλλον θα καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρω τη χρηματοδότηση. Επίσης κάναμε αλλαγές στην ε, υλοποίηση, για συγκεκριμένα στον κανονισμό υλοποίηση, Έτσι θα απλουστευθεί κάπω το έργο των κρατών μελών. πρέπει να εκπονηθεί έκθεση για την εμπειρία μας από το πρόγραμμα αυτό «Φρούτα στα σχολεία». Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τα τέλη του 2012. Και λόγω αυτών των προβλημάτων που είχαμε και με προβλήματα ελέγχου, γιατί θέλω να σας πω ότι σε σχέση με το πρόγραμμα για το γάλα, ουσιαστικά ακολουθήσαμε ως πρότυπο αυτό το σύστημα για το γάλα, με τα, την ε, διανομή γάλακτος στα σχολεία. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τόσο πρόβλημα λοιπόν, αφού ουσιαστικά αντιγράψαμε αν θέλετε ένα άλλο σύστημα, αλλά υπάρχουν ε, κάποια ε, ζητήματα διοικητικά και οι συνάδελφοί μας από τη Γενική Αρμόδια Γενική Διεύθυνση θα δουν τι διοικητικό άχθος προέκυψε και θα έχουμε και τη σχετική έκθεση. Ελπίζουμε μέχρι το καλοκαίρι. We have established a so-called stakeholder group. stakeholder group Επίσης, το Φεβρουάριο είχαμε μια συνάντηση της ομάδας εργασίας. Θα έχουμε και φέτος ε, στις 24 Μαρτίου μια συνάντηση αυτής της ε, διευρυμένης ομάδας ε, που την απαρτίζουν μπλεκόμενοι φορείς και άνθρωποι του management της διοίκησης από τα κράτη-μέλη. Επίσης θα συγκροτήσουμε μια επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνοντας κάποια επιστημονικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά επίσης ε, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών, θα προσπαθήσει να μοντελοποιήσει το πρόγραμμα αυτό ώστε να είναι πιο ορθολογικό και δράτω με τις ευκαιρίες για να σας πω ότι το πρόγραμμα Φρούτα στα σχολεία από μόνο του δεν αφορά τόσο πολύ το να ταΐσουμε φρούτα και λαχανικά τα παιδιά στα σχολεία. Είναι περιορισμένο το ποσό ε, των 90 σε σχέση με το τι μπορούμε να πετύχουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε όμως ε, είναι να ανοίξουμε την πόρτα στα λεγόμενα συνοδευτικά μέτρα, αυτό το μήλο, την ένα μήλο την εβδομάδα, αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, τα συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών, στα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα όπου σε συντονισμό με τον ακαδημαϊκό κόσμο, με κόσμο από την και Γεωργία κτλ. να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα για να δουν πώ μπορούν στα σχολεία στη διδακτέα ή στο πρόγραμμα σπουδών να εντάξουν την έννοια τη διατροφής, των τροφίμων, της γεωργίας, ε, του περιβάλλοντο κτλ. Έτσι τα παιδιά μας θα μπορέσουν να ωφεληθούν και να ξαναέλθουν σε επαφή με την Ήπεθρο, αυτό που έχει χαθεί στην πόλη, σχέση με την Ήπεθρο, με την Γεωργία. Προσπαθούμε επίσης να αυξήσουμε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά. Όταν, δηλαδή ακριβώς στη στιγμή που σχηματίζουν και διαμορφώνουν τις διατροφικές του συνήθειες θέλουμε να επηρεάσουμε σε αυτή την ηλικία τα παιδιά. Και θέλουμε βέβαια να κινητοποιήσουμε και την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, όχι μόνο από τα παιδιά, αλλά και από τους γονείς τους, ε, τα αδέλφια τους, ε, των παιδιών δηλαδή, ε, από τους εκπαιδευτικούς. Άρα θέλουμε και θα έχουμε, πιστεύουμε, ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα καλύψει ε, ένα ευρύτερο, μια ευρύτερη ομάδα στόχων. Μπορώ να πω λοιπόν προς το παρόν κύριε Πρόεδρε ότι το πρόγραμμα αυτό αποδίδει. Ε, πιστεύουμε ότι μπορεί βέβαια να ε, βελτιωθεί ιδίως ό,τι αφορά τα γραφειοκρατικά προβλήματα και έχουμε και αυτή την πτυχή της χρηματοδότησης που όπως είπα για κάποια κράτη-μέλη πραγματικά είναι ένα εμπόδιο και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρο. ευχαριστώ πολύ τον διευθυντή Χέλγκαρτ. Ο συνάδελφο Λαβία έχει ζητήσει το λόγο, ο Τζιωβάνι. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή, η Κομισιόν μας έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Αλλά στο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε 22 εκατομμύρια παιδιά υπέρβαρα και ένα, 1,5 εκατομμύριο παιδιά τα οποία είναι επικινδύνως υπέρβαρα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα του αυξημένου βάρους της παχυσαρκίας των παιδιών μας αφορά όλους. Θα πρέπει τουλάχιστον ε, να καταναλώνουν 450 γραμμάρια φρούτων και λαχανικών την ημέρα. η συγχρηματοδότηση αυτού του προγράμματος, η ανάγκη συγχρηματοδότησης έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην εφαρμογή του προγράμματος. Ορισμένες χώρες της Ένωσης έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα, άλλες όχι ή όχι στον ίδιο βαθμό. Έχει λοιπόν μία διακύμαση στην εφαρμογή το πρόγραμμα. Ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν πώς γίνεται στο κείμενο του κανονισμού έχουμε ένα χρηματοδοτικό όριο, ένα όριο χρηματοδότησης το οποίο δεν υπάρχει σε άλλα προγράμματα. 90 εκατομμύρια ευρώ το οποίο βεβαίως ε, περιορίζει τα περιθώρια λιγμού δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό άργησε να αναπτυχθεί, να ξεκινήσει. Ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν πώς γίνεται αυτές οι ομάδες εμπειρογνωμόνων που υποτίθεται θα υποστήριζαν και θα βοηθούσαν στην εδραίωση αυτού του προγράμματος από το 2009 δεν το έχουν ακόμα κάνει το 2011 και δεδομένο ότι ο κανονισμός λέει για τα συνοδευτικά μέτρα 1,3 εκατομμύρια ευρώ ε, και για να χρηματοδοτηθούν και οι αιτήσιε συναντήσει, ο συντονισμό μεταξύ των προγνωμών κλπ. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν ήδη γίνει, δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Όλα αυτά τα συνοδευτικά μέτρα είναι σημαντικά για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, για να γίνει ευκολότερη η υλοποίησή του. Σαφώς ε, από απόψεως υγείας ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Γιατί λοιπόν δεν έχει ακόμα πλήρως εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή για, τις, για ε, ε, ε, την υπερστατωμένη ανάλυση και τους προλαλήσαντες. Εγώ θυμάμαι το ξεκίνημα αυτού του προγράμματος και ε, μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ε, που μου έλεγαν τουλάχιστον στη Γερμανία είναι η συνεννόηση με τα διοικητικά εμπόδια. Ε, θα ήθελα να εξαλειφθούν όλα αυτά τα διοικητικά ή τα γραφειοκρατικά εμπόδια για να μπορέσει να γίνει πλήρωση η υλοποίηση. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα να ασχολούμαστε με το να τρώνε τα παιδιά περισσότερα φρούτα. Ε, είναι πολύ σημαντική βεβαίως ε, η διατροφή των παιδιών αλλά θα πρέπει να τα διαμορφώνουμε έτσι ώστε να εφαρμόζονται και εύκολα το πρόγραμμα είναι θαυμάσιο και μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Αλλά η διαχείριση του προγράμματος και τα διοικητικά προσκόμματα, τα, τα προσκόμματα στην υλοποίηση είναι ακόμα σημαντικά. Πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε όχι μόνο στη διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων αλλά και στην διευκόλυνση της εφαρμογής τους. υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και είναι πολύ σημαντική η εξάλληψη, τουλάχιστον η των πιο σημαντικών γραφειοκρατικών εμποδίων για να μπορέσει ε, το πρόγραμμα να αναπτυχθεί στρωτά. Ευχαριστώ. Ελίζαμπεθ και πάλι ο κύριος Σόλγκαρτ. Ευχαριστώ. Um, Πολύ σύντομα, επειδή τέθηκε το ερώτημα για το όριο της χρηματοδότησης των 19 ε, ε, νομίζω εκατομμυρίων ευρώ. α, αποφασίστηκε αυτό το κείμενο του κανονισμού πριν από τη συναπόφαση. Ίσως δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά έτσι έγινε. Τώρα, όσον αφορά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν, είπα ότι δημιουργήσαμε δύο ομάδες. Η μία περιλαμβάνει τους ενδιαφερόμενους του κλάδου, του τομέα και η άλλη είναι η ομάδα των επιγνωμόνων η πρώτη συνεδρίαση των, της ομάδος των stakeholders, των ενδιαφερομένων, ήδη έγινε ε, φέτος, ε, το Φεβρουάριο, και η συνάντηση των εμπειρογνωμών θα γίνει σύντομα. Όσον αφορά την ιστοσελίδα, ναι, δέχομαι την παρατήρηση, θα βελτιωθεί. Ε, εδώ πρέπει, έχουμε περιθώριο βελτίωσης και στο σχεδιασμό και στη λειτουργία της ιστοσελίδας. Για να είναι όσο το πιο εύκολη στη χρήση της, φιλική στο χρήστη. Επίσης, ε, όσον αφορά τώρα τα γραφειοκρατικά εμπόδια έπρεπε να γίνει μια εσωτερική διαδικασία υποβολής αιτήσεων, εξέτασης ε, των αιτήσεων και πολύ σύντομα, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα ποια ημερομηνία, αλλά όλο το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτό το πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι το ξεκίνησα εγώ και το υποστηρίζω ένθερμα αλλά μην ξεχνάμε ότι πάντοτε πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ εποπτείας, ελέγχου και ορθολογικής υλοποίησης. Πάντοτε υπάρχουν ε, διοικητικά και γραφειοκρατικά κολλήματα, αλλά προχωρούμε όσο μπορούμε καλύτερα και ταχύτερα. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, άλλοι ομιλητές, θα συνεχίσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μπορούμε, ωραία. Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομική πόρη για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Ο εισηγητής είναι Τζοβάνι Λαβία. Μετά από απόφαση Ε, για την προετοιμασία μιας ε, γνωμοδότησης θα ζητήσω από τον κύριο Λαβία να παρουσιάσει ε, την γνώμη των συντονιστών και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μέγκλε. Στη σύνταξη της γνωμοδότησης πρώτα απ' όλα επαναλαμβάνω το περιεχόμενο του σημειώματος που είχε σταλεί Εμείς θέλαμε να μην πρόκειται για μια απλή νομοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συμπληρώνουν πλέον την κοινωνική πολιτική. Στόχος μας δεν πρέπει να είναι μόνο παραγωγή, ποσότητα, ποιότητα, αλλά είναι διαφορετική πλέον η ποιότητα, αν θέλετε αγαθών που παράγει μεν ο αγρότης, αλλά για τα οποία δεν λαμβάνει καμία αντιστάθμιση και καμία αμοιβή. Για να υπάρξει λοιπόν μεταφορά πόρων προς ε, την Ήπεθρο πρέπει να είναι πιο οικολογική και κοινή γεωργική πολιτική. Αυτή η γεωργική πολιτική απαιτεί έναν προπολογισμό που να είναι τουλάχιστον ισότιμος με αυτόν που έχουμε σε αυτή την περίοδο προγραμματισμού. Δεν μπορεί να διανοούμαστε ότι με συμπληρωματικέ απαιτήσει που θα επιβαρύνουμε, τις οποίες θα επιβαρύνουμε τον ε, γεωργικό χώρο, του γεωργού, θα του δώσουμε και λιγότερου πόρου από ό,τι ως σήμερα προβλεπόταν. Στην έκθεση έχω υπογραμμίσει και άλλε δύο πτυχέ. Μία είναι αυτή της διάρκειας του πολιετούς πλαισίου προγραμματισμού. Διότι η πείρα μας τώρα, ιδίω στην ανάπτυξη της υπαίθρου, μας δείχνουν ότι σε μία περίοδο προγραμματισμού, πολύ συχνά τα πρώτα χρόνια του, προ της περίοδου ε, αρχή, αφοσιώνονται στην περίοδο έναρξης των προγραμμάτων, στο startup. Ενώ στη συνέχεια υπάρχει μια, ένας διαγωνισμός τρεξίματος για να προλάβουν οι διάφορες περιοχές τις δαπάνες και για να μην επιστρέψουν στους πόρους τους μη εκτελεσμένους τα ποσά. Εδώ λοιπόν για την ε, καλή χρήση, την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων που αποδίδονται στην ανάπτυξη τη Πέθρου, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Μια τρίτη πτυχή είναι αυτή που έχει να κάνει με τη διάρθρωση του προπολογισμού. Αυτό το έχει δει και η Επιτροπή για το, που είναι υπεύθυνη για τις νέες πολιτικές προκλήσεις και το πολιετές πλαίσιο προγραμματισμού για τους πόρους που αποδίδονται στα διάφορα κεφάλαια της Γεωργίας, είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο πυλώνα, εκεί θεωρώ ότι είναι εύστοχο να διατηρήσουμε μια διεύθυνση του υπολογισμού ανάλογη με αυτή που σήμερα έχουμε. Με ένα κεφάλαιο που να αφοσιώνεται συγκεκριμένα στην στήριξη της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εδώ θα σταματήσω και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω στις ερωτήσει που θα τεθούν. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον, στην κυρία Γκαρσία Περές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να πω ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος συμφωνούμε με τα σημεία που ανέφερε ο κύριος Λαβία τα οποία συμπεριλαμβάνει και στο σχέδιο γνωμοδότησής του. Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες του και η Επιτροπή μας έχει ήδη αποφανθεί στο πλαίσιο διαφόρων εκθέσεων σε σχέση με το τι χρειάζεται η κυνηγυρική πολιτική για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές που συζητούμε. Αυτό το οποίο ίσως ανησυχεί λίγο είναι αυτό το σκηνικό όταν από τη μια πλευρά έχουμε την ε, πιθανότητα του ενδεχόμενο μείωσης ε, των εισφορών των ε, κρατών μελών στον προπολογισμό με την εισαγωγή νέων πολιτικών. Δεν θα πρέπει για να μπορέσουμε να έχουμε νέες πολιτικές να διατηρήσουμε την πρικοδότηση του προπολογισμού. Πρέπει να γίνουν σημαντικέ κοινέ προσπάθειε, σημαντική δουλειά και τη Επιτροπή Γεωργία του Κοινοβουλίου ώστε να μπορέσουμε κι εμείς ε, να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα σε σχέση με την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Η σοσιαλιστική ομάδα έχει συγκροτήσει τις δικές της ομάδες εργασίας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών και έχουμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις ε, προτείνει. Νομίζω ότι αν όλοι πάμε προς την ίδια κατεύθυνση θα είναι εύκολο κατά την άποψή μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, γνωμοδοτήσει ε, ως προς τις εξής γραμμές, να διατηρήσουμε την προκοδότηση της ΚΑΠ που ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια μειώνεται ο προϋπολογισμός της και πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε και νέες προκλήσεις. Εξού και είναι απολύτως απαραίτητο τουλάχιστον να διατηρηθεί η τρέχουσα χρηματοδότηση και με τα ίδια χαρακτηριστικά και με τον ίδιο προγραμματισμό όπως μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε, Ράς, ο Τζόρτζ Λάιον. Ε, πρόεδρε, συνάδελφοι, να πω ότι σε γενικές γραμμές στηρίζω το σχέδιο έκθεσης που μας έχετε υποβάλει. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα συνοπτικό και πυκνό σε νόημα. Πηγαίνει στην ουσία του θέματος και είναι πολύ καλό να δούμε τα επίπεδα τη περίοδου προγραμματισμού στο 2013 για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Να το σκεφτούμε από τώρα λοιπόν και σωστά μιλάτε για τι επιπλέον περιβαλλοντικέ υπηρεσίε που δεν θα καλύπτουν στο μέλλον οι γεωργοί. Όπω ίσω κάνουν σε ένα βαθμό τώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίζουμε ότι χωρί τον δέοντα προπολογισμό δεν μπορούμε να πετύχουμε κάποιου από του στόχου που έχουμε θέσει σε προηγούμενε εκθέσει και που ενδεχομένω να επανελάβουμε σε μια από τι επόμενε εκθέσει μα με τον κύριο Ντέσλεγου χάρη. Χρειάζεται εδώ και ευελιξία, όπω σωστά λέτε, γιατί αν σκεφτούμε ότι η περίοδος προγραμματισμού ε, στο 2013 λήξει με, μια περίο μια, ένα ποσοστό εκτέλεσης 39,3% εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με περιπτώσεις κρίσεως, κρίσεων μάλλον, όπου θα υπάρξει έκτακτη ανάγκη παρέμβασης. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και στο πώς θα προχωρήσουμε, τι θα γίνει για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες κρίσεις, τι εργαλεία δημοσιονομικά θα έχουμε στα χέρια μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες έκτακτες ανάγκες. Ευχαριστούμε, Τζόρτζ. Ο κύριος Η κυρία Ρέιμερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η έκθεση σωστά εντοπίζει ότι πρέπει να θέσουμε στόχου μακροπρόθεσμου, αλλά πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί σε σχέση με όσα είπε ο κύριο Λάιον. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με του στόχου που θέτουμε, διότι εάν δεν έχουμε του απαραίτητου πόρου, δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα τη αγορά. Αυτό λοιπόν το μέσο είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για μας είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πρικοδότηση από την πλευρά του υπολογισμού, περισσότερου πόρου. Τι τελευταίε εβδομάδε είδαμε πόσο σημαντική είναι η προμήθεια και πρώτων υλών, για, ακόμη και για την πολιτική σταθερότητα μια χώρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος, προστασία στην παραγωγή των τροφίμων, γιατί η προστασία των ιδιών διατροφή πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά τη γεωργική παραγωγή. Δεν μπορούμε αυτό να το ξεχνάμε. Τα επόμενα χρόνια η παραγωγή των ιδιών διατροφή θα είναι ένα μέσο για να εγγυηθούμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στι περισσότερε χώρε. Έπειτα, περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη και περισσότερη μεταφορά τη έρευνα και ανάπτυξη προ τη Γεωργία. Και αυτά είναι πολύ σημαντικοί στόχοι. Ευχαριστούμε η κυρία Μαγκίνε. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λαβία για αυτήν την ε, πολύ εύστοχη έκθεση. Εδώ παρεμβαίνω για να συμφωνήσω με την κυρία Ρέμερ για την σημασία της παραγωγής τροφίμων. Στην ε, Ολομέλεια καλωσορίσαμε τη συζήτηση για τις τιμές των τροφίμων και μάλιστα στο μέσο της ημέρας στο Στρασβούργο. Συνήθως τα θέματα αυτά τα συζητάμε μεσάνυχτα εκεί. Η σημασία λοιπόν των τροφίμων είναι ζωτική και εδώ η πραγματικότητα επιβάλλει να προβλέψουμε και απαραίτητου πόρου από την πλευρά του προπολογισμού για τη γεωργική πολιτική. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία και αυτό όπω το υποστηρίζει η έκθεση. Και εδώ τον συσχετισμό με την έρευνα και τη μεταφορά γνώση θα την υποστηρίξω επίση προ την παραγωγή τροφίμων. Εάν δείτε την παράγραφο 5, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, λόγω των ε, πολλών στόχων που ε, προβλέπουμε να ε, λάβουμε υπόψη την ιεράρχηση και για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών και αυτό είναι σημαντικό, και στην παράγραφο 2. Η, τα πολλαπλά ζητήματα, όπω η περιβαλλοντική προστασία, η ζωική ε, ευζοία, και οι νέοι στόχοι με τους νέους πόρους που θα εξασφαλίσουμε στην ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε τον εισηγητή λοιπόν για αυτή την έκθεση και να πω ότι όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, εάν εδώ είμαστε ενωμένοι και ισχυροί ως Επιτροπή και προβάλλουμε την ανάγκη ενός ε, υψηλού προπολογισμού για την ε, Γεωργία, νομίζω θα έχουμε επιτελέσει κάποια πρόοδο. Ευχαριστούμε Μαρέιντ, ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με όσα προτείνει ο συνάδελφος Λαβίας στην έκθεσή του. Θεωρώ ότι η διάρθρωση του προπολογισμού έχει αυτή τη στιγμή ε, δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη ε, τις γεωργικές ανάγκες Πρέπει να είναι πιο ευέλικτο λοιπόν ο προπολογισμό, αλλά να προσέξουμε η πολλή ευελιξία να μην αποστραγγίξει τους πόρους της Γεωργίας προς άλλα λίματα, Διότι έχω την εντύπωση, γνωρίζοντας τα όσα συζητούνται και στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, ότι αυτή η τόσο επιδιωκόμενη ευελιξία μπορεί να γίνει ένα όχημα για να απομακρύνουμε πόρους και ποσά από τα όσα προορίζονται για την γεωργία. Σε, όσα, σε σχέση με όσα μόλις είπε η συνάδελφος Μαγκίνες, να πω ότι και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος είναι κάτι που εξηγεί το γιατί χρειαζόμαστε δαπάνες για τον γεωργικό προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τις ανάγκες του ευρωπαϊκού πληθυσμού, διότι η επιστημιστική ασφάλεια είναι ένα υψηλή ε, αξία αγαθό. Κάτι που συχνά το παραμελούμε. Ξεχνάμε ότι τα αγαθά αυτά παράγονται από μια ομάδα πολιτών, του γεωργού, οι οποίοι λίγο πολύ κερδίζουν τα μισά από όσα ο γενικότερο πληθυσμό. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν το εισόδημά του είναι δίκαιο. Είναι σωστό να παίρνουν τόσα λίγα. Και βεβαίω από την άλλη πρέπει να δικαιολογήσουμε και τι δαπάνε προ την Γεωργία. Όλη αυτή η συζήτηση ε, και σε σχέση με το περιβόητο cleaning πρέπει να γίνει με τρόπο πιο σαφή, διότι είναι πολλοί ο κόσμο που δεν καταλαβαίνει κατά πόσο γνωρίζουμε σωστά τι δαπάνε μα. Ευχαριστούμε ο κύριο Γκλάτενφελντερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ άριθμες οι μελέτες και οι συνεδριάσεις και οι συσκέψεις που γίνονται που γίνεται λόγος τελευταία για το γεγονός ότι η μέγιστη πρόκληση τα ερχόμενα χρόνια θα είναι τα προβλήματα της ενέργειας και η έλλειψη νερού και τροφίμων. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι προβληματισμοί είναι στοιχεία που τα γνωρίζουμε. Ήδη έχουμε τα πρώτα προειδοποιητικά σήματα, το τι συμβαίνει με την ενέργεια, τα τρόφιμα, είναι θέματα που τα γνωρίζουμε. Η επισητιστική λοιπόν ασφάλεια γίνεται ένα νέο ζήτημα που αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του ζητήματο αυτού, καλό θα ήταν να τοποθετηθούμε αποτελεσματικά ω Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι διακυμάνσει των τιμών. Ε, εδώ θα πρέπει η παρέμβαση που θα προβλέψουμε ή μάλλον το σύστημα παρεμβάσεων που θα προβλέψουμε με τα απαραίτητα αποθεματικά να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει παρέμβει στην αγορά των δημητριακών. Εκεί, πέραν των υψηλών τιμών που βλέπουμε σήμερα, θα ήταν σημαντικό να είχαμε και αποθέματα τα οποία θα πολλούσαμε σε συμφέρουσες τιμέ, πράγμα που θα μας επέτρεπε να πολλαπλασιάσουμε τις πηγές εσόδων για την κοινή γεωργική πολιτική. Όμως η έλλειψη παρέμβαση έχει προκαλέσει απώλειε για του ίδιου του παραγωγού και για του καταναλωτέ και τελικά ωφελήθηκαν μόνον οι εταιρείε, οι εμπορευόμενοι σε διεθνεί συναλλαγέ που αποφελούνται από τη διακίνηση αυτών των πρώτων υλών. Επίσης για την διαχείριση των υδάτων. Και εδώ θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερους πόρους προκειμένου να διευκολύνουμε την άρδευση και να προλάβουμε τα προβλήματα των πλημμυρών και των βροχοπτώσεων. Τώρα, για την ε, ενέργεια, το αν η Γεωργία είναι ο πιο σημαντικό χρήστη ενέργεια. Αυτό είναι μέρο τη λύση, όχι του προβλήματο. Διότι θα μπορούσε η Γεωργία να συμβάλλει στι προσπάθειε εξοικονόμηση ενέργεια, όπω λόγου χάρη με τη βιομάζα που παράγονται χάρη στι γεωργικέ δραστηριότητε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα από τα μεγαλύ... μια από τις σημαντικότερες πηγές ενέργειας και η γεωργία θα πρέπει να πρικοδοτηθεί με συγκεκριμένους υποχρεωτικούς ε, δημοσιονομικούς ε, σκοπούς και πόρους προκειμένου να επιτελέσει με επιτυχία αυτόν της το ρόλο και μετά το 2013. Ευχαριστούμε κύριε Γκράτενφέρντερ, ο κύριος Ανιώ και μετά ο κύριος Μποδέ. Πρόεδρε, ε, άγνιο ονομάζομαι και ίσως είναι λίγο δύσκολο να το δείτε από εκεί που κάθεστε, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λαβία. Για τις ε, προτάσεις που έκανε χωρίς να αναφέρει την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Τον ευχαριστώ ολόθερμα γι' αυτό. Γιατί πολλοί από εμά στο Ηνωμένο Βασίλειο που παράγουν ζαχαρότευλα, έχουμε χάσει ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματό μας λόγω του παγετού, του κρύου, του τσουκτουερού κρύου. Και παρόλα αυτά μας λένε ότι πρέπει να αυξήσουμε και το αποτύπωμα του άνθρακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που είπατε. Οι δύο λοιπόν μεγάλες προκλήσεις της ε, πολιτικής μας είναι η, η πάγια καταβολή στους ε, παραγωγούς η οποία σιγά σιγά διαφεύγει από τα χέρια των ε, παραγωγών και πηγαίνει στα χέρια των μεγάλων ιδιοκτητών γης. Η άλλη μεγάλη πρόκληση που έχουμε είναι ότι τα κονδύλια του δεύτερου πυλώνα θα πρέπει να δαπανηθούν λογικά ε, και να μην πάνε χαμένα, όπως έχει γίνει τόσες φορές στο παρελθόν. Ευχαριστώ κύριε Άγνιο, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Μπούβε. Ναι. Κάποια σημεία τα οποία δεν έχουν ε, αναφερθεί, ε, να τα προσθέσω λοιπόν. Πρώτον, κάτι που πρέπει να επενθυμίσουμε, είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε, είναι το εξή. Αν θέλουμε πράγματι να είναι επαρκή ο προϋπολογισμός, θα πρέπει τα σχέδια που θα προωθήσουν στον τομέα της ε, γεωργίας ε, να είναι θεμητά. Αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε αυτά τα σχέδια. Θα κάνουμε και τη συζήτηση μετά για αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρώτα απ' όλα οι Ευρωπαίοι πολίτες χρηματοδοτούν μέσω, τους φόρους μέσω των φόρων που πληρώνουν αυτά τα σχέδια, άρα θα πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους. Δύο σημεία θέλω να υπογραμμίσω τα οποία μέχρι σήμερα ακόμη δεν έχουν θυγεί. Παραδείγματο χάρη, επανεξισορρόπηση δημητριακά κρέας. Σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα δημόσιας ιδιωτικής αποθήκευσης δημητριακών σιτηρών σε περίπτωση κρίσεων σαν αυτή που βιώσαμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει μια νέα γραμμή να εφαρμοστεί, γιατί όλα τα προηγούμενα εργαλεία τα έχει καταστρέψει η Κομισιόν. Και σήμερα που βιώνουμε αυτή την κρίση, ούτε η Κομισιόν ούτε τα κράτη έχουν τα μέσα στη διάθεσή τους για να προωθήσουν την αποθήκευση σιτηρών, να υπάρχει μια τυποποιημένη τιμή τους και για, το ζωικό κεφάλαιο. Δεύτερον, σημαντικό και για τη γεωργία και για την κατανάλωση, είναι το θέμα του όλο και σημαντικότερου ελέγχου των θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία. ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Η ΕΦΣΑ δεν έχει οικονομικούς πόρους για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στις αξιολογήσεις που κάνει. Δύο δυνατότητες λοιπόν έχουμε. Ή στηρίζουμε την ΕΦΣΑ με δημόσια κονδύλια και τα, τη στηρίζει και η Κομισιόν ή την ΕΦΣΑ τη στηρίζει τη στηρίζουν ε, επιχειρήσεις. Βλέποντας όμως τα σκάνδαλα σήμερα, σύγκρουση συμφερόντων, σχέσεις με επιχειρήσει. νομίζω ότι θα πρέπει στον προβληματισμό που κάνουμε να προβλέψουμε την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την ενίσχυση του προπολογισμού τη. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και να προχωρήσουμε σε αυτό στη συζήτηση που θα κάνουμε. Ευχαριστούμε, Ζε. Ο κύριος Σιλβέστρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ να εκφράσω την μεγάλη μου εκτίμηση για το σχέδιο έκθεση που μα προτείνει ο συνάδελφο ε, Λαβία. Όχι γιατί μόνο κάθεται δίπλα μου στα έδρανα και είμαστε και από το ίδιο κόμμα και από την ίδια χώρα, δεν είναι μόνο για αυτό που τον εκτιμώ, αλλά γιατί πραγματικά εκφράζει κάτι που όλοι συμμεριζόμαστε. Ουσιαστικά έχει συμπυκνώσει τις βασικές ιδέες για το θέμα αυτό με, ένα, με πολύ σωστούς συλλογισμούς. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποσκοπήσουμε και ένα σημαντικό στοιχείο, την προοδευτική μείωση των ποσοστώσεων, του ποσοστού που αφιερώνεται ε, στην ΚΑΠ, στον προπολογισμό τον ευρωπαϊκό από 85% να περνάει στο 75% με 3% επίσης ε, από το 2013 και μετά. Αυτό ε, για συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτό δείχνει ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε την κοινή αγροτική πολιτική. Ίσως και εμείς είμαστε πολύ παθιασμένοι με μια συζήτηση που αυτή τη στιγμή όμως απασχολεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να εξεύρει μια εξίσωση. Να αποδείξει δηλαδή ότι οι πόροι της γεωργίας αποδίδονται σε μια ε, πολιτική η οποία έχει να κάνει με την επιβίωση και την παραγωγή. Πρέπει να δείξουμε τόλμη από δική μα πλευρά. Δηλαδή να τοποθετηθούμε κατά τον αντίθετο τρόπο. Να αποδείξουμε ότι τα ποσά που αποδίδονται στην γεωργία εξασφαλίζουν το κοινό συμφέρον όλων, όχι μόνο των γεωργών. Είναι χρήματα που θέλουν να εξασφαλίσουν την επιστημιστική επάρκεια, ε, την καλή κατάσταση της υπαίθρου και των ε, επαρχιών και την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών προϊόντων στην διεθνή μάλιστα αγορά. Και αυτό είναι σημαντικό μερίδιο τη ε, συνολική μα οικονομική δραστηριότητα και τη αγορά μα. Δυστυχώ όμω δεν καταφέρνουμε πάντοτε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή εισοδήματα για του γεωργού. Διότι τελικά με την εξίσωση αυτή που λέει ότι οι πόροι που αποδίδονται στην ε, γεωργία έχει να κάνει με μια, με μια πολιτική μόνο ε, για την παραγωγή, καταλήγει στο να μην επωφελούνται παρκώ οι γεωργοί από τα ποσά που αποδίδονται στην ΚΑΠ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να μην επιδοθούμε σε διανοητικέ ε, ασκήσει, αλλά να είμαστε πρακτικοί στο σχεδιασμό τη έκθεση αυτή. Δεν μπορούμε να μην διατηρήσουμε αυτό το ποσοστό του προπολογισμού για την ΚΑΠ από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Θα πρέπει να το υπερασπιστούμε με μεγάλη τόλμη, με μεγάλη αποφασιστικότητα και να αποδείξουμε τη χρησιμότητα και την ευστοχία των πόρων που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει στην κοινή αγροτική πολιτική. Έτσι λοιπόν, συμμερίζομαι πλήρω όχι μόνο τι θέσει του σχεδίου έκθεση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το επέβαλε ο εισηγητή. Είναι πολύ συνοπτικό, σαφή και εύστοχο. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο Γενικός, ε, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Μέγκλε για τα σχόλιά του και μετά ο κύριος Λαβία για να κλείσουμε. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω καταρχάς ότι το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Λαβία αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τη συζήτηση που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ε, μελλοντικές προοπτικές και τις πολιτικές προκλήσεις μετά το 2013. Έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αγροτική πολιτική μετά το 2013 και φιλοδοξία μας είναι επίσης μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες γιατί και το πρόγραμμα ε, του Επιτρόπου μου διότι θα το συζητήσουμε αυτό στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης αλλά πιστεύω ότι θα αναφερθεί στις ε, προκλήσεις που έχουν επισημανθεί στην Ατζέντα 2020 ε, στις προκλήσεις του περιβάλλοντος επίσης και Πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να ε, είναι η χαρακτηριστική, να είναι δυνατή η συμβολή μας από την πλευρά του αγροτικού τομέα. Ε, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν όλες αυτές οι θαυμάσιες ιδέες αν τα κονδύλια μειωθούν είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε τους παραγωγούς να ακολουθήσουν την ε, κατεμά σωστή κατεύθυνση εάν ταυτόχρονα επιβάλλουμε περικοπές. Γι' αυτό είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την, ε, στο σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Λαβία, ο οποίος λέει ότι τα κονδύλια, οι για την αγροτική πολιτική μετά το 2013 πρέπει να είναι επαρκή, έτσι ώστε να μπορέσει η ΚΑΠ να επιτελέσει το ρόλο της. Αυτό το οποίο ε, τονίζει το σχέδιο γνωμοδότησης είναι η ευελιξία. Βεβαίως, η ευελιξία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και θα είναι και μετά το 2013. Όμως να προσέξουμε διότι η ευελιξία μπορεί να ακολουθήσει διάφορες κατευθύνσεις. Θα πρέπει η το προτινόμενο στοιχείο ευελιξίας να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί και σε μέτρα εκτός αγροτικής πολιτικής και να μην εφαρμοστεί η ευελιξία σε μέτρα τα οποία θα διακυβεύσουν τους κοινούς στόχους μας για την αγροτική πολιτική. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, το στοιχείο που θέλω να τονίσω στο σχέδιο γνωμοδότησης είναι ότι θέλει να διατηρήσει την κοινή αγροτική πολιτική υπό ένα κεφάλαιο για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προπτικές. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, διότι η αγροτική πολιτική δεν είναι ένα θέμα το οποίο να έχει μια αριστερή πτυχή, μια δεξιά πτυχή, αλλά είναι ένα ενιαίο σύνολο και ως ενιαίο σύνολο πρέπει να τη δούμε όταν μιλάμε για μέτρα ε, της αγοράς, για την παγκόσμια οικονομία και παγκόσμια στοιχεία. Γι' αυτό πρέπει να διατηρήσουμε οπωσδήποτε τους δύο πυλώνες ως έχουν και μαζί ενοποιημένα να θεωρήσουμε την πολιτική αυτή στον προϋπολογισμό. Πιστεύω και επαναλαμβάνω αυτά που είπα στην αρχή ότι το σχέδιο γνωμοδότησης αποτελεί μια εξαιρετική βάση συζήτησης, ε, συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάσινση ε, τη συζήτηση στον αγροτικό τομέα και στο μέλλον της ΚΑΠ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γενικό Διευθυντή και τώρα να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. δηλαδή, Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, για όποιου θέλουν να υποβάλουν τροπολογίε, είναι στι 2 Μαρτίου το μεσημέρι στι 12. Μέχρι μεθαύριο ουσιαστικά στι 12. Τζοβάνι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την συζήτηση που είχαμε. Να ξεκινήσω με ένα αστείο. Τόσα χρόνια ασχοληθήκαμε με σύνθεση διαφορετικών ιδεών. Όποιος όμως καλείται να σχεδιάσει μια έκθεση ξέρει ότι υπάρχει και ο περιορισμός στους χαρακτήρες. Άρα υπάρχει ε, περιορισμός από τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου στη σύνταξη μιας έκθεσης ε, για τους λόγους της, για τους σκοπούς της μετάφρασης. Είναι αναγκαστικό να είναι κανείς συνοπτικός στη σύνταξη μιας έκθεσης τέλος πάντων. Και αυτό τι δέσμευση, αυτό ο φραγμό δεν ισχύει για τι τροπολογίε. Οπότε σκέφτηκα κάτι να το ε, συμπληρώσω από τι τροπολογίε, προσθέτοντα κάποιου χαρακτήρε στο συνολικό όριο. Τέλο πάντων, νομίζω ότι ακούσαμε πολλά σοβαρά στοιχεία από την ε, συζήτηση και πολλέ επικοδομητικέ παρατηρήσει. Θα πω, χωρί να μπω στι λεπτομέρειε, ότι νομίζω το σημαντικότερο ζήτημα είναι αυτό τη ευελιξία. Γιατί? Γιατί όλοι γνωρίζετε ότι με τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχει ξεκινήσει μια διαφιλονικία μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής. Για το θέμα αυτό ακριβώς, της ευελιξίας, η συνθήκη της Λισαβόνας θα προέβλεπε βάση των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου κάτω του 0,03% και εφόσον υπάρχει θέμα επιλογής μεταξύ λιμάτων του προπολογισμού, εκεί να αποφασίζει ομόφωνα το Συμβούλιο. Αυτό φαίνεται αρκετά δύσκολο όμως να συμβεί. Είναι λοιπόν σαφές ότι η χρηματοδότηση της κοινή αγροτικής πολιτικής συσχετίζεται αναπόφευτα με ένα ζήτημα που είναι ευρύτερο, το θέμα της ευελιξίας στο πλαίσιο του κοινοτικού προπολογισμού. Αυτό είναι ένα ζήτημα που η Επιτροπή Σούρε θα πρέπει να εξετάσει, μαζί με την ομάδα εργασίας που ακριβώς ασχολείται με το δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να βρεθεί μια λύση που να επιτρέπει να προχωρήσουμε και να επιτρέπει να είναι εφικτή και μεταφορά των πόρων μεταξύ κεφαλαίων του προπολογισμού. Κατά τα άλλα, είναι επίσης σαφές ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει ως στόχο να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την παραγωγή τροφίμων για την κοινότητα, την ευρωπαϊκή κοινότητα. Αυτό που συμβαίνει τώρα, ειδικά στην, περίοδο, στην περιοχή μάλλον της Μεσογείου, δεν είναι παρά ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με μεγάλες χώρες παραγωγούς δημητριακών, όπως η Ρωσία, που θέλει να παρατείνει την ε, μείωση των εξαγωγών για να διασφαλίσει την δική της επισητιστική επάρκεια. Θα πρέπει λοιπόν εδώ την κοινή αγροτική πολιτική να την δούμε συνολικά πέραν των ε, πρόσθετων στόχων που έχουμε θέσει στα πλαίσια αυτή τη γενική μεταρρύθμιση, πρέπει να παραμείνουν στου πρωτογενεί στόχου. Παραγωγή τροφίμων, επάρκεια στην προμήθεια τροφίμων στον Ευρωπαίο πολίτη. Σε αυτό ακριβώ το πλαίσιο, που ούτω ή άλλω θα το αναπτύξουμε περιττέρω στα πλαίσια τη έκθεση DES για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία που μπορούμε να προσθέσουμε στην όλη συζήτηση. Έγινε λόγος και για έρευνα και ανάπτυξη. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο διεθνέ ε, πολιτικό σκηνικό είναι σημαντικό στα πλαίσια της νέας ε, κοινή αγροτικής πολιτικής να δώσουμε ένα πρωταρχικό ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παρεμβληθεί αυτό στην έκθεσή μας ώστε να υποδείξουμε μια κατεύθυνση προς αυτήν την πορεία και επίσης για τους θεμετούς στόχους, για το πόσο είναι θεμετή μάλλον η ΚΑΠ. Ε, σίγουρα πρέπει να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως είπε και ο Ζωζεμποβέ, ότι αυτήν την πολιτική τη χρειάζονται και είναι θεμητή. Ελπίζω στη δική σας συμβολή λοιπόν ε, και την άμεση, συζητώντα μαζί μου, και με τις τροπολογίες σας, προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της έκθεσης. Και κάτι τελευταίο, ο Ζωζέμποβε αναφέρθηκε στα υγειονομικά προβλήματα, στη χρηματοδότηση της ΕΦΣΑ επίσης. Αυτό έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελείως διαφορετικό κεφάλαιο. Εκεί προφανώς θα μπορούσαμε να επανέλθουμε όταν συζητήσουμε για τον προπολογισμό. Εκεί θα πρέπει να εξακριβώσουμε τι βήματα μπορούμε να προβλέψουμε ώστε να δώσουμε μεγαλύτερο έλεγχο για τα θέματα αυτά στους ευρωπαϊκούς Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους και σας ευχαριστώ και παραμένω στη διάθεσή σας για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής και υπό το φως των παρατηρήσεων της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Τζοβάνι Λαβία. Εγώ ευχαριστώ προφανώ όλου του συναδέλφου. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο. Το πλέον σημαντικό τη ημερήσια διάταξη. Η κοινή γεωργική πολιτική στον ορίζοντα του 2020. Εξέταση του σχεδίου έκθεση. Συνάδελφοι, εδώ δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω τη σημασία του θέματο αυτού και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ντε, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του, να σας πω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το στάδιο αυτό. Και πόσο σημαντικό επίσης είναι να είμαστε ενωμένοι εδώ. Όσο πιο συμπαγής είναι η τοποθέτησή μας, τόσο περισσότερο θα επηρεάσουμε τις επιλογές που θα κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή στις νομοθετικές της επιλογές. Με αυτήν λοιπόν την προκατακτική παρατήρηση δίνω το λόγο στον κύριο Ντες, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του και στο μεταξύ να ευχαριστήσω για την ε, παρουσία, την παρουσία του τον κύριο Φράνκο Κυριακό, ε, ε, εισηγητή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και εντωμεταξύ ας δώσω το λόγο στον κύριο Ντες ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι της Κομισιόν και παρόντες ακροατές, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα την έκθεση για την κοινή γεωργική πολιτική με χρονικό ορίζοντα μετά το 2013, χρονικό το 2020. Μετά από την έκθεση του Γκέρο Κλάιεν και μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν, είναι σειρά του Κοινοβουλίου και πάλι να παρουσιάσει τις απόψεις του και να εκφράσει τις επιθυμίες του. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Επίτροπο για τις ε, ανακοινώσεις του και αναφέρουμε τις προτάσεις του και αναφέρουμε σε πολλά μέρη της έκθεσής μου στις προτάσεις του. Όπως επίσης και σε πολλά στοιχεία της έκθεσης του κυρίου Λάιεν. Ευχαριστώ τον κύριο Λάιεν για όλες τις προσπάθειές του. Στην έκθεση αναφέρουμε σε πολλές λεπτομέρειες, αυτό ίσως σας ξαφνιάσει, δεδομένου ότι με την συναπόφαση που έχει τώρα το Κοινοβούλιο βάσει της Λισαβόνας θα πρέπει να αναλάβει έναν ισχυρότερο ρόλο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να παρουσιάσει τη δική του θέση για να μπορέσουμε να αντιποκριθούμε σωστά στις νέες αυτές ευθύνε. και αρμοδιότητες. Βεβαίως το Κοινοβούλιο πρέπει να εργαστεί με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για να βρούμε κοινή θέση στα θέματα της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Η βάση της έκθεσής μου λέει ότι η κοινή πολιτική, η γεωργική πολιτική πρέπει να γίνει απλούστερη και, και σαφέστερη. Πιο απλή για όλους τους εμπλεκόμενους, τους παραγωγούς, ε, τους εμπορευόμενους, ε, τους διαχειριστές ο στόχος μας πρέπει να είναι η απλούστευση. Αυτό είναι το υπερσμόν ένα συμπέρασμα της έκθεσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει μετά το 2013 να έχουμε μία αξιόπιστη, ε, εφαρμόσιμη ε, και υγιή ε, όσον αφορά την χρηματοδότηση κοινή γεωργική πολιτική. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την κοινή γεωργική πολιτική γιατί καταρχάς προς όφελος των παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την επισητιστική επάρκεια του πληθυσμού μας που φτάνουν περίπου το μισό δισεκατομμύριο. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε τα τρόφιμα που χρειάζεται ο πληθυσμός μας, αλλά και να εκμεταλλευτούμε με σοφροσύνη τους πόρους που έχουμε. Η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της έκθεσή μου. Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους χρειαζόμαστε, έτσι όπως το είπε ήδη ο George Lane και η ανακοίνωση της Κομισιόν, δύο πυλώνες, αρχιτεκτονική δύο πυλώνων. Χρειαζόμαστε μία σαφή δομή, ξεκάθαρη δομή αυτών των πυλώνων, χωρίς να υπάρχουν επικαλύψεις και παρανοήσεις που οδηγούν στην περαιτέρω αύξηση της γραφειοκρατίας. Μία ισχυρή, ένας ισχυρός πρώτος πυλώνας είναι λίγαν σημαντικός για την επίτευξη των υψηλών κοινωνικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την επίτευξη όλων των κοινωνικών ε, στόχων για τη μείωση των κινδύνων των ε, παραγωγών μας και για την ομαλή εξέλιξη των κινδύνων από εξωτερικές ε, πηγές αλλά και βεβαίως πάντοτε για την επίτευξη της επιστημιστικής επάρκειας. Ακούσαμε σήμερα τις ε, δυσκολίες που υπάρχουν ε, στη ζάχαρη. Παραδείγματο χάρη, ορισμένα προϊόντα αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν έλλειψη. Πριν από 20 χρόνια η παραγωγή ζαχαρωτών και γλυκών είπαν ότι υπάρχει αρκετή ζάχαρη στον κόσμο, ρυθμίστε επιτέλους τις ανομαλίες της αγοράς, μπορούμε να εισάγουμε από άλλα μέρη του κόσμου και να λύσουμε τα προβλήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα πολλές φορές αντί να διευκολύνονται δυσκολεύουν. Επίσης υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα οι διαφορές αυτές έχουν οξυνθεί, όχι εξομαλυνθεί. Η κοινή γεωργική πολιτική θα είναι σωστή και θα υλοποιηθεί σωστά εάν εκμεταλλευτούμε καλύτερα τα κοινά στοιχεία και όχι τις διαφορές μας. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να εργαστούμε προς μία υφόρο γεωργική ανάπτυξη και για την εξάλληψη των ελλημάτων όπου αυτά παρουσιάζονται. Ε, θα πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε ικανοποιικά τις πληρωμές στον πρώτο πυλώνα. Το σύνθημά μας πρέπει να είναι όχι περαιτέρω επιβαρύνσεις για τους παραγωγούς και την ε, δίκηση, τη διαχείριση και τη δίκηση. Το καθεστώς όλο πρέπει να απλουστευθεί, να γίνει πιο δίκαιο, πιο ευέλικτο, πιο επικεντρωμένο σε συγκεκριμένους στόχους. Αυτά θα μπορέσουμε να τα επιτύχουμε οδεύοντας προς το δεύτερο πυλώνα χωρίς να ε, δημιουργηθούν στρεβλώσεις και ζημιές. Κύριε Πρόεδρε, στις 2 ε, Μαΐου από ό,τι ξέρω θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και μετά στην Ολομέλεια. Έχουμε λοιπόν, όπως βλέπετε, αρκετό περιθώριο να συζητήσουμε ενδελεχώς όλα τα στοιχεία της έκθεσης. Ε, θα ήθελα ακόμα να πω γιατί ε, θεωρώ ότι ο δεύτερος πυλώνας είναι τόσο σημαντικός. Έχω μία ανοιχτή προσέγγιση. Όταν κάποιος, εάν κάποιος μου προτείνει ότι θα πρέπει και να εξαλειφθεί η γραφειοκρατία και στον πρώτο πυλώνα ε, θα πω ότι ναι, εντάξει, αλλά δεν έχω ακούσει προτάσεις για την μείωση ή την εξάλληψη της γραφειοκρατίας στον πρώτο πυλώνα. Και δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό ε, με όλες αυτές τις διαφορές που υπάρχουν στους παραγωγούς μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν παραγωγοί που λαμβάνουν 50 ε, ή 600 ευρώ και ένα μικρό ποσοστό παραγωγών ε, ε, λαμβάνουν 15 ευρώ ή 180 ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αποφασίσουμε ίδιες τιμές αναφοράς και ίδιες τιμές αποθεματοποίησης. Δεν μπορούν να υπάρχουν αυτές οι τεράστιες διαφορές. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το σύστημα μπορεί να απλουστευτεί μέσω του δεύτερου πυλώνα. Διαπιστώνω στις συζητήσεις που κάνουμε ότι πολλοί παραγωγοί ακόμα έχουν στο μυαλό τους τα, λεφτά του πρώτου πυλώνα και πιστεύουν ότι τα λεφτά του πρώτου πυλώνα είναι σίγουρα λεφτά ενώ του δεύτερου είναι, δεν είναι σίγουρα, είναι, τα αμφισβητούν. Εμείς ε, θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη η ίδια προσέγγιση ε, των ενδιαφερομένων και στους δύο πυλώνες. Δηλαδή να υπάρχει βεβαιότητα για, τα, για τις πιστώσεις και μέσω του πρώτου και μέσω του δεύτερου πυλώνα. Ε, πιστεύω ότι το, το η υλοποίηση του συστήματος δεν εφαρμόζεται ενιαία στα κράτη-μέλη, δεν έχω όμως ακόμα βρει λύση για τον ορισμό του μικρού παραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό διαφέρει τόσο πολύ το, το καθεστώς ε, στην εφαρμογή όλων των μέτρων στους μικρούς παραγωγούς. Εγώ πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν ένα, ένα ποσό, ε, ορισμένες πιστώσεις από τον πρώτο πυλώνα για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους μικρούς παραγωγούς έτσι όπως τους ορίζουν εν πάση περιπτώσει. Αλλά ενιαία λύση του ορισμού δεν έχω βρει. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ενδεχομένως να υπάρξει ένα ε, υποχρεωτικό ποσοστό διάθεσης πιστώσεων για τους μικρούς. Επίσης για τους νέους παραγωγούς και, και αυτό μας απασχολεί. Ξέρω ότι πολλοί νέοι παραγωγοί έχουν προβλήματα σημαντικά σε ευρωπαϊκά κράτη ε, να λάβουν, ε, να δανειστούν, ε, να, να πάρουν πιστώσεις και δάνεια τα οποία χρειάζονται για τη μονάδα τους. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε και αυτό το θέμα να το καλύψουμε στο δεύτερο πυλώνα. Πιστεύω επίσης ότι το σύστημα ως έχει δημιουργεί ε, Διακρίσει σε ορισμένε περιφέρειες ε, όσο, όπως έχει σήμερα στο δεύτερο πυλώνα και πρέπει να διορθωθεί. Μπορούμε μέτρα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ των κρατών μελών να τα εξομαλύνουμε στο δεύτερο πυλώνα. Εάν δούμε, δεν πιστεύω Πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε διάφορες βαθμίδες στο δεύτερο πυλώνα. Δηλαδή να διασπάσουμε αυτόν τον άξονα και να δημιουργήσουμε διάφορα μπλοκ, τα οποία μπλοκ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσω της ε, χρηματοδότησης με υποχρεωτικές πιστώσεις σε παραγωγούς οι οποίοι τις δικαιούνται από τον πρώτο πυλώνα. Το ένα δεύτερο μπλοκ του δεύτερου πυλώνα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να διαθέσουμε πιστώσεις για περιβαλλοντικά μέτρα που θέλουν να εφαρμόσουν οι παραγωγοί. Ε, ας πούμε 75% χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση, 25% συγχρηματοδότηση από το κράτος μέλος. Και όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, και πάλι εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε εκτός ορισμένων εξαιρέσεων ένα μπλοκ συγχρηματοδότησης 50-50. Ε, 50 ευρωπαϊκά, 50 εθνικά πιστώσεις, κονδύλια. Αυτή η συγχρηματοδότηση λοιπόν ε, πιστεύω ότι μπορεί να χειριστούμε ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Για τα μέσα εφαρμογής ε, στην αγορά πιστεύω ότι αυτά τα, αυτές οι πράξεις, αυτά τα μέσα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα θα πρέπει να διατηρηθούν έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις κρίσεων και να τα εμπλουτίσουμε σε περίπτωση που διαπιστώνουμε πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στις αγορές. Συμφωνώ με τον Αντιπρόεδρό μας και συμφωνώ και το έχω γράψει και σε επιστολή ότι θα πρέπει να σκεφτούμε εάν επανέλθουμε στο παλαιότερο σύστημα των ελάχιστων αποθεμάτων, εάν θέλουμε να περιορίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα των, ε, της κερδοσκοπίας θα πρέπει να σκεφτούμε εάν θέλουμε, εάν πρέπει σε ορισμένα χρονικά διαστήματα να, υπάρχει, να υπάρχουν ορισμένες μίνιμουμ ποσότητες σε απόθεμα. Ε, θα μπορέσουμε Λοιπόν, να συνδέσουμε αυτό το θέμα και την αντόπιση αυτού του προβλήματος με τα γενικότερα προγράμματα της Ευρώπης 2020. Πρόσφατα διάβασα μία έξεση προγνωμόνων ότι από τις 10 καλύτερες ε, ε, αγροτικές περιοχές που παρουσιάζουν τις καλύτερες ε, γεωργικές προοπτικές στην Ευρώπη. Τρεις από τις δέκα αυτές βρίσκονται στη δική μου περιφέρεια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ε, στη Γερμανία έχουν πραγματικά εξελιχθεί πολύ σημαντικά και σε πολλές περιφέρειες επιτυχώς οι αγροτικές δομές. Ελπίζω να μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και οι άλλες χώρες και περιφέρειες που ακόμα μειονεκτούν. Περιμένω με ανυπομονησία και με μεγάλο ενδιαφέρον τις συζητήσεις που θα κάνουμε, τις προτάσεις που θα ακούσω. Όσοι με ξέρουν γνωρίζουν ότι είμαι πρόθυμος ε, να κάνω συμβιβασμούς και ε, πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε μία έντονη και ενδιαφέρουσα συζήτηση τις επόμενες μέρες και εβδομάδες και ότι στο τέλος με μεγάλη πλειοψηφία θα καταφέρουμε να περάσουμε ε, μια έκθεση του Κοινοβουλίου η οποία θα βοηθήσει και θα προσφέρει πολλές ιδέες στον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και περιμένω να ακούσω ε, και, προσβλέπω με μεγάλη χαρά στην περαιτέρω συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστούμε. Οπωσδήποτε θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. 20 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Πρώτα απ' όλα όμως θα δώσω το λόγο στο Φράνκο Κυρίακο διότι όπως βλέπεις Φράγκο, έχουμε λίγο χρόνο. Θα σου ζητήσω λοιπόν να είσαι ο πιο συνοπτικός γίνεται. Εισηγητής της ε, Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ε, διότι σήμερα, ε, όπως είπα και προηγουμένως, ψηφίστηκε το ίδιο θέμα στην ε, Υποεπιτροπή ΝΑΤ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε στη συνεδρίασή σας. Όπως σωστά είπατε κι εσείς, το ειδικό τμήμα που είναι επιφορτισμένο με θέματα γεωργίας, ανάπτυξης υπαίθρου και περιβάλλοντος στην Επιτροπή μας, ψήφισε και ενέκρινε την έκθεση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η τελική συζήτηση θα γίνει στην Ολομέλειά μας στις 15 Μαρτίου. Εποφελούμε εδώ λοιπόν για να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ντες, ε, για τις εργασίες που έχει κάνει ως σήμερα και επισήμως ε, θα ξανασυζητήσουμε την δική σας την έκθεση με τα μέλη της δικής μας Επιτροπής. Εγώ είμαι Γεωργός. Είμαι μέλος της ομάδας 2 και εκπροσωπώ τους εργαζομένους. Ε, άρα είμαι μέλος, μέρος του κόσμου αυτού. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ βασική αρμοδιότητα και στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι να εναρμόσει τα συμφέροντα των γεωργών με τις ανάγκες των πολιτών καθότι παράγουν ε, τρόφιμα και πρώτης ανάγκης ήδη. Θα πρέπει να του εξασφαλίσουμε εισόδημα αξιοπρεπέ σε όλου του γεωργού, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή ο γεωργό, ο δραστήριο γεωργός θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγωγής, να μπορεί να εμπορεύεται τα προϊόντα του και πολλές φορές μάλιστα πουλώντας τα άμεσα σε τοπικές αγορές. Εμείς ως Επιτροπή συμφωνούμε ότι χρειάζεται κάπινγκ όπως προτάθηκε από τον Επίτροπο στην σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής. Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όχι μόνο εξαιτία της ε, εντατικότητας της μισθωτής ε, ε, εργασίας, αλλά και στην μη αμοιβόμενη εργασία του Γεωργού. Θεωρώ λοιπόν ότι στη χρηματοδότησή μας θα πρέπει να προβλέπεται και μια κοινωνική δικαιολόγηση και να φανεί και προς τους πολίτες γιατί χρησιμοποιούνται οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν έχουμε τονίσει Τρει βασικούς στόχους. Το περιβάλλον, τις ανάγκες των γεωργών και την εργασία. Ο γεωργό δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πρόστο στοιχείο και να υπολογίζεται το κάπινγκ ή για να ε, μπορεί να γίνεται ένα στοιχείο στη σύγκριση της ζωικής ε, ε, Είναι ανθρώπινο το κεφάλαιο εδώ. Μιλάμε για 18 εκατομμύρια εργαζομένους της Ευρώπης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της γεωργίας. Και υπάρχουν άλλα 4 εκατομμύρια που δεν μπορούν να εντοπιστούν, δεν ε, έχουν κάποια συγκεκριμένη σύμβαση και σε πολλές ε, περιοχές της Ευρώπης, σε πολλά κράτη είναι ε, παράνομοι, παρανόμως διαμένοντες. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια προσέγγιση ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει στον αγροτικό τομέα την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, όπω είπε ο κ. Ντέ και συμφωνούμε, και να συνεισφέρει στη βελτίωση των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων, δηλαδή ασφάλεια των εργαζομένων, ε, δίκαιη αμοιβή και συμμόρφωση με τις κοινωνικές ρήτρες. Τελευταία παρατήρηση και κλείνω. Η Επιτροπή μας θεωρεί ότι είναι αδύνατο, όπως σωστά υπόθηκε, να πραγματοποιηθεί αποτελεσματική μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής μετά το 2013, εάν δεν υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση για τη διάσταση που έχει να κάνει με τη διάρθρωση του υπολογισμού. Αυτό είναι κεντρικής σημασία σημείο. Για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθούν στόχοι, εργαλεία και δημοσιονομικά μέσα. Να εντοπιστούν όλα αυτά στην συγκεκριμένη έκθεση προκειμένου να βρεθεί σωστή ισορροπία. Πρόεδρε, να θυμίσω εδώ ότι το άνοιγμα τη αγορά θα οδηγήσει σε εντατικοποίηση του ε, ανταγωνισμού, σε αύξηση των τιμών και θα υπάρξουν και πολλέ εισαγωγέ commodities κοινών αγαθών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνουμε συνεχώ υπόψη την πραγματικότητα των αγορών. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα υπάρχοντα μέσα στην, ε, σε ανάγκη σταθεροποίηση Τη ίδια τη αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Φράγκο Κυριακό. Τώρα ξεκινούμε την συζήτηση. Να δώσω πρώτα το λόγο στου εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Και μετά σε όλους του υπόλοιπου. Προ στιγμήν έχουν εγγραφεί 23 αγορητέ. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε κάπως. Ε, Λουίς θα ξεκινήσεις εσύ. Ο κύριος Καπούλα Σάντος. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ συνοπτικός και όσο γίνεται αντικειμενικός. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντες για το έργο του. Ε, ήταν εντατική εργασία τον τελευταίο καιρό, τον παρακολουθήσαμε και ήταν και αρκετά δυσχερή κάποιε φορέ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν εδώ τονίζοντα κάποιε πτυχέ που θεωρώ θετικέ στην έκθεση. Ο συνάδελφο Ντε ακολουθεί την έκθεση Lions σε κάποιε αδρέ γραμμέ και κάποιε από τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτές πρέπει και εμείς να συμφωνήσουμε. Έτσι λοιπόν θετική αποτίμηση για την ενίσχυση της γεωργικής πολιτικής, ενίσχυση του πρωτοπυλώνα, επανακατυποποίηση κάποιων στοιχείων, διανομή δικαιότερη και πιο ισότιμη των πόρων μεταξύ των κατώμελών και των ίδιων των γεωργών. Προτάσεις απλούστευσης, υπεράσπιση ενός καθεστώτος πληρωμών με κοινωνική μέρημνα και ανάλογα με την επιφάνεια και σε μια μεταδοτική μεταβατική περίοδο εκτό από έκτακτε περιπτώσει. Και το ιστορικό κριτήριο για την απονομή βοήθεια στου γεωργού θα πρέπει να συζητηθεί σοβαρά. Αυτέ είναι οι θετικές πτυχές. Κατά τα άλλα, και εδώ, για να είμαι πολύ ειλικρινή στην κριτική μου και πολύ πραγματιστή, θεωρώ από την άλλη ότι η έκθεση αυτή είναι αρκετά ασαφή. Δεν είναι ακριβή σε κάποιε πτυχέ για τι οποίε το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτή τη φάση δεν μπορεί παρά να τοποθετηθεί παρόλα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάπω ασαφή και άσυνεπή η τοποθέτηση για την κεντρική ιδέα του κειμένου. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω συνοπτικά τι εννοώ η έκθεση του κυρίου Ντες προτείνει μια εθελούσια βάση για την πληρωμή ε, των ε, ενισχύσεων στους γεωργούς. Γιατί εθελοντική. Από τη στιγμή που θα ορίσουμε μια πολιτική με κοινού κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζεται και πραγματικός ανταγωνισμός. Ε, ο συνάδελφος Ντες δεν κάνει καμία πρόταση για τον ορισμό της ε, ενεργής γεωργίας. Εδώ δεν μπορούμε απλώς να ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίζει τα κριτήρια. Έχουμε υποχρέωση μέσω μιας έκθεσης να υποβάλουμε και εμείς μια πρόταση. Το η ομάδα των σοσιαλιστών έχει ιδέες εδώ να παρουσιάσει και θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Ε, το η έκθεση DES μιλάει για την δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ενισχύσεων και προτείνει το κάθε κάτω μέλο να λαμβάνει λιγότερο από τα δύο τρίτα του μέσου όρου των πληρώμων που έχουν δοθεί ω τώρα. Μα για ποιο μέσο όρο μιλάμε όμω, τον τωρινό μέσο όρο, τον μέσο όρο που προκύπτει μετά από την εφαρμογή των νέων κριτηρίων αυτό είναι κεντρική σημασία στοιχείο. Είναι πολύ ε, σημαντικό να αποσαφινιστεί στην συγκεκριμένη έκθεση. Επίση, ο συνάδελφο Ντε προτείνει την πρόσθετη κάλυψη κινδύνων. Όμω δεν λέει πιανών κινδύνων. Ε, στο σημείο 33 μιλά για πρόσθετη λοιπόν κάλυψη, αλλά μετά στο εδάφιο 40 μιλά για απόλυτη απόρριψη του συστήματο ευρωπαϊκών ασφαλιών. Ε, αυτό μου φαίνεται αρκετά αντιφατικό. Επίση, ω προ την στο σημείο 52 ως προς την ανάπτυξη καλή πραγματικά ε, σε συγχρηματοδότηση. Μια πτυχή που οδηγεί σε επανακριτικοποίηση της ΚΑΠ, της κοινή γεωργικής πολιτικής. Από τη μια λοιπόν είναι κατά της επανακρατικοποίηση, αλλά στο σημείο 35 και 52 καλεί σε συγχρηματοδότηση ε, ε, από τα εθνικά κράτη. Επίσης, όπως είπε ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή, εδώ ε, η διάσταση της ε, απασχόλησης και της εργασίας που ανέφερε εκείνος δεν υπάρχει καθόλου σε αυτή την έκθεση. Ε, το κριτήριο της απασχόλησιμότητας, της απασχόλησης, είναι μεγάλη παράληψη να μην ε, προβλεφθεί εδώ πέρα. Και άφησα τελευταίο το ζήτημα που θεωρώ ότι είναι το πιο αμφιλεγόμενο στην έκθεση αυτή, το σημείο 22, το πιο διαφιλονικούμενο αν θέλετε. Εδώ Νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι τελείω συγκεχημένη και τελείω ε, ε, αντιφατική σε σχέση με τι αρχέ απλούστευση που η έκθεση προτίθεται να εισαγάγει. Εδώ δεν μπορούμε να προτείνουμε πληρωμέ 100% χρηματοδοτούμενε από το δεύτερο πυλώνα όταν μπορούν να προκύψουν από τον πρώτο. Άρα είναι αδύνατο να συμφωνήσουμε ως σοσιαλιστές. Εδώ και, κάποιου μήνε, εδώ και κάποιους μήνες ε, θέλουμε ενίσχυση του πρώτου πυλώνα με παρόμοια μέτρα, μέτρα αγροτικά και περιβαλλοντικά που θα έχουν περάσει στο δεύτερο πυλώνα και θα έχουν προστατευτεί και εξασφαλιστεί πολύ καλύτερα εκεί. Το είπε πριν από λίγα λεπτά. Τα λόγια του ήταν. Οι Γεωργοί θεωρούν τον πρώτο πυλώνα σίγουρα κονδύλια και τελείω ε, αβέβαια αυτά του δεύτερου. Άρα τα των αγροτικών περιβαλλοντικών ε, στοιχείων, ε, γιατί να μην περάσουν στον πρώτο πυλώνα, ώστε να υπάρξει μια μετατόπιση και να εξασφαλίσουμε τις ανάγκες των μεν και των δε. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη αυτού του στόχου, μπορούμε να αναζητήσουμε την κατάλληλη έκφραση για όλε αυτέ τι προτάσει και ελπίζω ότι η σοσιαλιστική ομάδα θα καταφέρει να κάνει τη φωνή της να ακουστεί. Δεν θέλω τώρα να περάσουμε σε μια συζήτηση μεταξύ των δυο μας για την όλη έκθεση. Νομίζω θα μπορούσαμε να σας φέρουμε θετικά στην σύνταξή της. Ευχαριστούμε ο κύριος Λάιον. Ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον Άλμπερτ Ντες για την σκληρή εργασία που έκανε στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Κατέβαλε έντονες προσπάθειες να συζητήσει με όλους τους ενδιαφερόμενους και δι' ε, με προσώπους της δικής μου ομάδας και μου προσωπικά Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις για τις, ε, τις, θέσεις, τις θέσεις που έχει εκφράσει στην έκθεσή του. Η ιδέα του για απλούστευση νομίζω δεν χωράει καμία αμφισβήτηση, είναι πάρα πολύ καλή. Επίσης η δίκαιη κατανομή πόρων, επίσης πολύ σωστή. Επίσης με ικανοποιεί το αίτημά του, οι πληρωμές να πηγαίνουν κατευθείαν και μόνον στους παραγωγούς. Ίσως θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα τον ορισμό όσον αφορά το capping και αυτό με ικανοποιεί και αυτό το δέχουμε. Υπάρχουν ορισμένες πτυχές της έκθεσης που με ανησυχούν και είχαμε την ευκαιρία να τις συζητήσουμε μέσα στην ομάδα μου. Το άρθρο 68 και στην παράγραφο 15 αναφέρεται στην ε, κατάρριση ορισμένων ενισχύσεων για τον γαλακτοκομικό τομέα και αναφέρεται και στη διάθεση πόρων του άρθρου 68 του κανονισμού για γάλα, πρόβατα, θυλάζουσες, αγελάδες κλπ. Θα ήθελα λοιπόν να έχω περισσότερες διευκρινήσεις για τις παραγράφους 15 και 16 των προτάσεων του. Ε, η μεγαλύτερη μου ανησυχία αναφέρεται στο θέμα της δίκαιης κατανομής της δικαιοσύνης, ε, της, του θεμητού αναφέρεται και στους δύο πυλώνες, στον πρώτο και στο δεύτερο, στο θέμα της ε, δικαιοσύνης, της, ε, ε, της δίκαιας κατανομής, της δίκαιης αντιμετώπισης και αναφέρεται επίσης ότι αυτό το στοιχείο του δίκαιου θα πρέπει να αντανακλά το 67% των άμεσων πληρωμών, 65% των άμεσων πληρωμών ε, που και στο 27% του μέσου όρου των άμεσων πληρωμών που κατά τους υπολογισμούς μου είναι 127 ευρώ που σημαίνει ότι μόνο τρία κράτη-μέλη θα ε, χαίρουν αυτού του Πλεονεκτήματο. Το μερίδιο των εξόδων προβλέπεται να μειωθεί από σχεδόν 75% σε 39% ε, της ε, πολιτικής και πιστεύω ότι με τις άμεσες ε, πληρωμές αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που μου δημιουργεί ανησυχίες. Και στην παράγραφο 22 των προτάσεών του αναφέρω αναφέρεται σε ένα, στην υλοποίηση ενός μοντέλου πιο απλού για τις άμεσες πληρωμές. Πιστεύω άμα εξετάσετε αυτή την παράγραφο το αυτό που προτείνει μάλλον είναι πιο περίπλοκο και όχι πιο απλό διότι ορισμένα κράτη-μέλη λέει πρόταση να μεταφερθούν κονδύλια από την πρώτο πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα, μετά θα έχουμε έναν κατάλογο μέτρων στο δεύτερο πυλώνα και αν δεν εμπίπτουν σε αυτό κατάλογο θα, τα χρήματα θα ξαναπάνε πίσω στον πρώτο πυλώνα. Ε, σε ορισμένα κράτη-μέλη οι πληρωμές γίνονται μέσω της μεταφοράς από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα σε άλλα κράτη-μέλη οι πληρωμές γίνονται μέσω άμεσων πληρωμών υπάρχουν λοιπόν δύο ροές χρηματοδότησης εάν λοιπόν ε, δεν τηρηθούν αυτές οι διαδικασίες πληρωμών θα επιβληθούν κυρώσεις και οι παραγωγοί θα χάσουν χρήματα τα οποία δικαιούνται. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ακριβώς ε, τι είναι αυτό το σύστημα που προτείνει στην παράγραφο 22. Πιστεύω ότι είναι πιο περίπλοκο από αυτό που έχουμε σήμερα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν περισσότερες ε, εξηγήσεις, περισσότερες διευκρινήσεις για το 22. Όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρους, ε, αναφέρεται σε ορισμένε περιφέρειες ε, προτεραιότητος, αλλά δεν αναφέρεται ακριβώς στην, ε, στις προτεραιότητες της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι προτεραιότητος μέσα στα πλαίσια της Ατζέντα 2020 πρέπει να καταλάβουμε, να έχουμε σαφή εικόνα ποιες περιφέρειες θα είναι ο στόχος μας και τι μέτρα θα εφαρμόσουμε εκεί προς όφελος ε, των παραγών και της κοινωνίας γενικώ. Ευχαριστούμε, Τζόρτζ. Ο κύριος Νίκολσον. Thank you very much, uh, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την ευκαιρία προσυζήτηση αυτής της έκθεσης. Πρέπει να αναγνωρίσω το έργο του κυρίου Ντες. Έχει βάλει ορισμένες νέες ιδέες και θα πρέπει να τις αναλύσουμε και να τις συζητήσουμε. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες πρωτοβουλίες τις οποίες έχει εδώ αναφέρει ο κύριος Ντες, έχει περιλάβει στην έκθεσή του και με χαρά θα τη συζητήσουμε. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να δουλέψουμε ως ένα σώμα, ως μία επιτροπή για να, μας, για να μπορέσουμε να, μας, να αυξήσουμε και το κύρος μας και να μας πάρουν στα σοβαρά. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη ευθύνη και πρέπει όλοι να συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Η απλούστευση την θέλουμε, τη χρειαζόμαστε. Μιλάμε ε, επιμακρών για την απλούστευση, αλλά δεν νομίζω να έχουμε επιτύχει και πολλά μέχρι τώρα πρέπει να απλουστεύσουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν και να είναι και απλουστευμένα ήδη αυτά τα, τα νέα στοιχεία. Δεν είναι απλό έργο αυτό. Ε, η απλούστευση μιας τεράστιας γραφειοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο για να μπορέσει να λειτουργήσει και να, το σύστημα και να έχουμε και τον έλεγχο του συστήματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι ε, η εμπιστοσύνη, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλα κραταμέλια, στη δική μου χώρα, αν καταργηθεί το, η άμεση πληρωμή η, η μία και μόνον πληρωμή στον παραγωγό δεν έχει καμία σημασία αν είσαι μικρή ή μεγάλη μικρή ή μεγάλη μονάδα. Εάν καταργηθεί αυτή η καταβολή θα καταστραφεί η βάση του γεωργικού τομέα της κονιακής ε, δομής και επιχείρησης. Θα διαλυθεί. Ευελιξία, επίσης, ευελιξία συμφωνώ. Ε, ευελιξία στον αφορά την ε, περιφερειακή ή εθνική εφαρμογή των μέτρων. Επίσης, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε, να φορέσουμε ένα κουστούμι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε, έχουμε διαφορές μεγάλες, ε, τοπικές, εθνικές και δεν μπορούμε όλα να τα κάνουμε ενιαία και ομοιόμορφα. Επίσης, με, με ανησυχεί η, η συγχρηματοδότηση δεν λέω ότι το κράτος έθνος ε, δεν θα πρέπει να έχει την ευελιξία και τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσει ειδικά του μέτρα, αλλά εάν προχωρήσουμε στην υποχρεωτική συγχρηματοδότηση, ή εάν η συγχρηματοδότηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, άλλα ωφέλη θα έχει μία δέσμη παραγωγών και άλλα ωφέλη θα έχει μία άλλη ομάδα παραγωγών και θα δούμε τα κονδύλια για την ανάπτυξη της υπένθρου στη δική μου χώρα δεν θα εφαρμοστούν τόσο καλά και δεν θα έχουμε τέτοια πλανεκτήματα όσο σε άλλες χώρες. Πολλές φορές η παραγωγή μου με ρωτάνε «Μα τι είναι αυτά που κάνετε» και τους λέω δίκιο να παραπονιέστε, ε, μπορεί να ε, είναι υποχρεωτική η χρηματοδότηση, αλλά εμείς από την εθνικής πλευρά δεν έχουμε τα λεφτά να τη σεβαστούμε» και να τηρήσουμε τα μέτρα αυτά. Καταλαβαίνω γιατί Όσον αφορά τους ορισμούς του παραγωγού, του παραγωγού ενδράση, ε, δεν ξέρω, καταλαβαίνω γιατί ο εισηγητής, ο συντάκτης της έκθεσης δεν προχώρησε σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα των ορισμών. Είναι σαν το κάπινγκ. Από τη στιγμή που ανοίγεις ε, το κουτί της Πανδώρας για όλες τις ερμηνείες και διευρύνεις έναν ορισμό τα, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Ε, βλέπω ε, Περιμένω λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον να δω τι θα φέρει αυτή η συζήτηση και πού θα καταλήξουμε. Λοιπόν, είπαμε ορισμοί, δύσκολο θέμα και ορισμένες ακόμα παρατηρήσεις. Χρειάζομαι περιττέρω διευκρινήσεις για αυτήν την ιδέα της εθνικής ασφάλειας έναντι ρίσκων, έναντι κινδύνων. Ασφάλεια έναντι κινδύνων. Ε, το, θέλω να ξέρω περισσότερα τι είναι αυτό, τι προτείνεται, τι ιδέα είναι αυτή και τι περιλαμβάνει. Πριν κρίνω, Επίσης χρειάζεται να υποστηρίξουμε αυτό το δίχτυ ασφαλείας ε, ε, ιδίως σε περιόδους κρίσης των αγορών, όταν η αγορά δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Γενικά όμως πιστεύω ότι η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να εργάζεται προς όφελος εκείνων που παράγουν τρόφιμα για την εξασφάλιση της επισητιστικής επάρκειας. Ε, βλέπουμε τι προβλήματα δημιουργούνται όταν δεν υπάρχει επάρκεια. Ε, και επίσης πρέπει να έχουμε μια ε, καλύτερη, μια διευκρίνηση γιατί είναι καλύτερα να μεταφέρουμε πιστώσεις από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 και μετά ξανά επιστροφή στον πυλώνα 1. Εγώ φοβούμαι ότι περισσότερη γραφειοκρατία θα επιβληθεί με αυτήν την προτινόμενη ιδέα παρά λιγότερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, James. Ο κύριος Όσλινγκ. Θα ήθελα και εγώ, λέει ο κύριος ε, Όσλινγκ, να ευχαριστήσω τον κύριο Ντες που ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο έργο κάποιο τεχνικό πρόβλημα στα ακουστικά. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να συμβάλλουμε και εμείς στην έκθεση αυτή ώστε να είναι τόσο καλή για να περάσει από το σώμα. Ε, πολλά θέματα τίθενται εδώ προς συζήτηση και πρέπει να τα συζητήσουμε λεπτομερώς. Καταρχάς συμφωνούμε στους δύο πυλώνες, στις δύο στήλες. Ε, ρωτώ όμως ε, γιατί ο συντάκτης λαμβάνει υπόψη, του δέχεται τις δύο στήλε, αλλά μετά αρχίζει τη, τη, τη γυμναστική της μεταφοράς κονδυλίων από εδώ και από εκεί. Ε, νομίζω ότι όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος με την έκθεση του χρειαζόμαστε μία το πρασίνισμα όλης της γεωργικής πολιτικής και γι' αυτό νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο, στην πρώτη στήλη. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να, ε, συντάξ, να προτείνουμε μέτρα ε, τα οποία θα ενισχύσουν ε, την πρώτη στήλη παραδείγματος χάρη σε συγκεκριμένα προϊόντα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και τους μηχανισμούς ελέγχου ιδιαίτερα σε θέματα. Πολλαπλή συμμόρφωση. Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η ενίσχυση των μικρών παραγωγών αλλά υπόθηκε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε εμάς τις πληρωμές στους μικρούς παραγωγούς αλλά μόνο όταν δεν στρεβλώνονται οι γενικές ε, αγροτικές δομές. Ε, εάν λοιπόν ε, ψηφίσουμε για μέτρα υποστήριξης των μικρών παραγωγών τα οποία όμως δεν εμποδίζουν τη μεταρρύθμιση, μεταρρυθμιστικές πτυχές δεν μπορεί να είναι σωστό αυτό. Θέλουμε και μεταρρύθμιση και ενίσχυση εν συνεχεία το διάστημα προσαρμογής ε, στις μεταρρυθμιστικές ε, προτάσεις. Ναι, βεβαίως έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική που πρέπει να τη δεχτούν ειλικρινά όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά τα προτινόμενα μέτρα για την επιβολή της δικαιοσύνης, της δίκαιης κατανομής, μιας δίκαιης πολιτικής και απόλυτα θεμητής προς όλους, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, πρέπει να σκεφτούμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το μέσο της αγοράς εργασίας. Παραδείγματος χάρη να λάβουμε υπόψη στην κατανομή των πιστώσεων της θέσης εργασίας. Δεν έχει υποθεί τίποτα σχετικό με αυτό. Πιστεύω ότι η αγορά εργασίας με τη δίκαιη κατανομή των πιστώσεων είναι αλληλένδετα. Συμφωνούμε στο άρθρο 68 ότι πρέπει να διατηρηθεί, ναι σωστά, ωραία. Επίσης, συμφωνούμε στην πρόσβαση της αγοράς ε, αλλά αυτό θα, αυτό πρέπει να ισχύσει και για τις ζωοτροφές ε, που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε ενδιαφέρον τη συζήτηση από αυτού, όχι μόνο επιστημιστική, επάρκεια, τρόφιμα κλπ, αλλά και ζωοτροφές εγώ θα ήθελα η έκθεση αυτή να ανταποκρίνεται περισσότερο στις απορίες που έχουν οι πολίτες μας, δηλαδή τι δαπανούμε και τι επιτυγχάνουμε, δηλαδή τη σχέση κόστους-οφέλους της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, δεν το γλιτώνουμε και να το αντιμετωπίσουμε δυναμικά και φιλόδοξα έτσι ώστε επιτέλους να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι του σώματος να συμφωνήσουν σε μια κοινή γεωργική πολιτική. Και τώρα προφανώς θα δώσω το λόγο στους υπολείπους συναδέλφους. Με τους συντονιστές ήμουν πιο ελαστικός, αλλά επειδή είναι 20 εγγεγραμμένοι, παρακαλώ θα συγκρατηθείτε όσο μπορείτε περισσότερο. Κύριε Παπαστάμκο. Πρόεδρε, ε, η αντικειμενική ανάγνωση της ε, έκθεσης του κυρίου Ντες οδηγεί σε συγκλήσεις και αποκλήσεις. Και διαβλέπω μάλιστα ότι οι συγκλήσεις ε, και οι αποκλήσεις θα συναντήσουν, θα κινηθούν σε διακομματική ε, βάση εδώ μέσα. Κάνω μια πρόβλεψη. Πέρα δηλαδή από το ΕΛΚ, πέρα από τους αριστές, πέρα από όλες τις ομάδες. Ε, θεωρώ πολύ θετικά, στοιχεία μεταξύ άλλων τη διατήρηση του προπολογισμού για τη Γεωργία μετά το 2013 τουλάχιστον στο ισχύον επίπεδο, ασφαλώς την εναντίωση στην επαναθνικοποίηση της ΚΑΠ και στη διατήρηση χρηματοδότηση των άμεσων πληρωμών αποκλειστικά από τον προπολογισμό της Ένωσης, η διατήρηση της αρχιτεκτονικής των δύο πυλώνων και την απλοποίηση εφαρμογής της ΚΑΠ προς όφελος των γεωργών, οι άμεσες πληρωμές είναι απαραίτητε για την ασφάλιση του γεωργικού συντήματο και για την αντιστάθμιση του υψηλού κόστου συμμόρφωσης με αυστηρά πρότυπα και την παροχή δημοσίων αγαθών τα οποία δεν διασφαλίζει η αγορά. Πάντως, ε, θα πρέπει να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των άμεσων ισχύσεων, ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκή μεταβατική περίοδο κάτι που είχε ο κ. Δε σε ένα ε, πρώτο σχέδιο τη έκθεση του. Διαφορετικά, οι κοινωνικονομικές επιπτώσεις θα είναι οξύτατες σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι δεν θα πρέπει να οριστεί ενιαία καταποκοπήν άμεση πληρωμή flat rate σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κρίσιμο παραμένει ε, λοιπόν να αναδείξουμε αντικειμενικά κριτήρια, το είπε και ο κ. Χόισλινγκ αυτό, για την κατανομή των άμεσων πληρωμών οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών. Χρειαζόμαστε δύο τελευταίες παρατηρήσεις, περισσότερο αποτελεσματικά και ευέλικτα μέτρα αγοράς. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή των ισιών των μέτρων αγοράς υπήρξε η ανεπαρκής. Τέλος, ό,τι αφορά το greening dimension, το πρασίνισμα, πιστεύω ότι πρέπει να επιλεγεί αποτελεσματικός αλλά και απλούστερος τρόπος δηλαδή ένας τρόπος που θα γιάται και τους αντίστοιχους πόρους υπέρ των παραγωγών. Αυτές είναι, αυτή είναι συνοπτικά μια πρώτη πρίμα φάτσιε ανάγνωση σε πολύ σύντομο χρόνο της έκθεσης του καλού συναδέλφου του κ. Ντες τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινώς για την ε, συμβολή του ε, και για το πρώτο αποτύπωμα των σκέψεών του σε αυτό εδώ το κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιώργος. Ευχαριστούμε Γιώργο. Η κυρία Γέγκλε. Το κύριο Ντόρφμαν μετά. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und zuerst einen herzlichen Dank an Albert, der sich mit seinem Bericht sehr, sehr viel Mühe. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Άλμπερτ πραγματικός έχει φέρει πέρα σε εδώ ένα τετάνιο έργο. Μελετώντας την έκθεση αυτή και συζητώντας για την κοινή γεωργική πολιτική στο μέλλον, δεν πρέπει να ξεχνούμε το εξής. Τι έχει προηγηθεί. Η έκθεση Λάιον, η έκθεση Παπαστάμκου για το διεθνές ε, εμπόριο. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη όταν μιλούμε για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Στο παρελθόν δεν είχε τόση σημασία για μας φαίνεται αυτό το θέμα, τώρα όμως έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Εάν λοιπόν δεν υπάρξουν αρκετοί πόροι, δεν θα υπάρξει κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητε στήριξη, γι' αυτό υπάρχουν και πολλέ ερωτήσει. Το σημείο 22 είναι μάλλον ένα από τα πιο δύσχεροι, τα πιο ακαθόδη. Δεν συμφωνούμε φυσικά πάντα, όμω εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Επίτροπο όταν αποδίδει Μάλλον δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον Επίτροπο όταν ε, προτείνει ένα ευρώ για το πρασίνισμα το λεγόμενο, το greening. Εδώ, μέσω από το δεύτερο πυλώνα, κάποια κράτη-μέλη κάνουν πολύ περισσότερα και κάποια άλλοι πολύ λιγότερα. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν του δεύτερου πυλώνα. Επίσης έχει ακουστεί η ιδέα να προβλεφθούν πόροι πολύ σημαντικότερη για τον πρώτο πυλώνα. Όμως εδώ πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Αν τα μέτρα του πρασινίσματος δεν περάσουν στο πρώτο πυλώνα, δεν θα καλύπτονται. Εδώ λοιπόν χρειάζεται έλεγχος. Λόγω χάρη στο δικό μου το κρατήδιο, το δικό μου land, είναι πολλά τα, μέτρα που έχουν ληφθεί. Ε, για το greening ακριβώς, για το πρασίνισμα, για την ε, οικολογική συνιστόσα. Ε, Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλύτερα να είναι υποχρεωτικά τα μέτρα αυτά και δεσμευτικά ε, και χωρίς χρησιμοποιηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα διάφορα είδη οποροκυπευτικών, φρούτα και λαχανικά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε άλλε χώρε. Δείτε τι γίνεται στο νότο τη Ισπανία. Είναι πολύ σημαντικό. Εάν θέλουμε να έχουμε πραγματικό greening, πρασινισμά, να το φέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα παρακαλώ λοιπόν θερμά να το έχετε αυτό συνεχώ κατά νου. Χρειάζονται παραχωρήσει, αλλά πρέπει να βρούμε και ένα στόχο τέτοιον, ώστε στο τέλο να μπορεί να γίνει και αποδεκτή έκθεση. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντόρφμαν, αλλά έχουμε ακόμη 17 εγγεγραμμένου και πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε. Θέλουμε και λίγο χρόνο για τους συντονιστές. Προσπαθείτε λοιπόν να συγκρατηθείτε παρακαλώ. Έρμπερτ. Και μετά ο κ. Μποβέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας ακολουθήσω στις συμβουλές σας. Εμείς ε, Εμεί, αν θέλετε, έχουμε επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην οικολογική διάσταση, στο λεγόμενο greening. Υπάρχουν σαφώ και άλλα σημαντικά όμω ζητήματα για το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν ε, πρώτα-πρώτα να δούμε τι συμβαίνει, τι κάνουμε τώρα για το greening. Μετά θα σκεφτούμε ποια θα είναι τα γεωργικά πριν για το περιβάλλον και θα δούμε και τι πόροι υπάρχουν στη διάθεσή μα. Θα σκεφτούμε επίση τι κάνουν οι μεν και τι οι δε, ποιοι κάνουν πολλά και ποιοι λιγότερα. Κάποιοι θα πανούν ένα 20% και άλλοι πολύ λιγότερο για τα προγράμματα ακριβώ περιβαλλοντικού χαρακτήρα που έχουν σχέση με τη γεωργία. Άρα πρέπει τα μέτρα του πρασινίσματος να υλοποιούνται και από τα κράτη-μέλη που για την ώρα έχουν μείνει σε χαμηλά επίπεδα. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και το εξής. Τα χρήματα θα πρέπει στον προπολογισμό να συμπεριλαμβάνονται στα σωστά σημεία, στα σωστά λήματα. Σίγουρα υπάρχουν απαιτήσει ιστορικού χαρακτήρα που επιβάλλονται από τις παραδόσεις ή τις συνήθειε. αλλα Αλλά κάποια κράτη-μέλη που βρεσκόντουσαν σε μειονεκτική θέση εργάστηκαν σκληρά και τώρα συνεχίζουν να λαμβάνουν πάρα πολλά παρόλο που έχουν επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δίκαιο. η καλλιέργεια δημητριακών λόγου χάρη που μας δίνει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία. Είναι λογικό αυτό, είναι λογικό να μην γίνονται επενδύσεις στο μέλλον των νεαρών γεωργών. Αυτά είναι για μένα κεντρική σημασία ζητήματα και ερωτήματα. Νομίζω ότι εξήλυσα τα δύο λεπτά, δεν έχω χρόνο να κάνω πολλές περι... περαιτέρω παρατηρήσεις, όμως Επιτρέψτε μου να πω για του μικρού γεωργού. Δεν ξέρω αν το θέμα είναι να πρέπει να πάρουν περισσότερα μικροί γεωργοί σε σχέση με του άλλου. Χρειάζονται όμω μέτρα για να του ελαφρύνουμε από τα γραφειοκρατικά του άχθη. Κύριε Μποβέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντες, πράγματι είχαμε την έκθεση στη γλώσσα μας τη μητρική, αλλά πολύ λίγο πριν την πήραμε στη γλώσσα μας, άρα ε, μπορώ να κάνω μια γενική ανάλυση επί της ουσίας και επί της μορφής. Καταρχάς, ό,τι αφορά τη μορφή, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό η έκθεση να διαρθρωθεί για να είναι κατανοητή, παίρνοντας το θέμα της παραγωγής, της κατανάλωσης και των γεωργών, σε αυτούς τους τρεις άξονες. Μόνο έτσι νομίζω ε, μάλλον έτσι γράφτηκε η συνθήκη τη Ρώμης, με αυτού του τρει άξους, τα τρία θέματα και έτσι καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι στόχοι τη κοινή γεωργική πολιτική. και θέλουμε έτσι να έχει συνέπεια, συνεκτικότητα το σχέδιο αυτό και να αντιστοιχεί με τι βάσει τη κοινή γεωργική πολιτική όταν ξεκίνησε το 1958. Είναι θέμα μορφής αλλά έχει και ουσία από πίσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι προκλήσει. Ε, δύο προκλήσει νομίζω αναφέρονται και είναι σημαντικό να τις επισημάνουμε. Πρώτη, ανακατανομή των ενισχύσεων. Πράγματι σήμερα είναι άδικη η κατανομή. Το αναγνωρίζουν όλοι, το αναγνωρίζει και η Κομισιόν. Σήμερα οι μισοί αγρότες δεν παίρνουν ενισχύσεις. Αν δει κανείς σήμερα, για παράδειγμα, ε, τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους, χείριου κρέατος ή πουλερικών που δεν έχουν καν έσοδα σχεδόν γιατί ανεβαίνει τιμή των πρώτων υλών. Δεν μπορούμε να τους στηρίξουμε αυτούς τους κτηνοτρόφους ε, γιατί δεν συμμετέχουν, δεν αποτελούν τμήμα αυτών που έχουν πρόσβαση στις ενισχύσεις. Άρα ανακατανομή ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ανακατανομή σε όλους τους αγρότες και μεταξύ των χωρών. Και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, το θέμα του περιορισμού των ενισχύσεων ε, ε, με ένα συγκεκριμένο πλαφόν, επίσης νομίζω ότι δημιουργεί ένα θέμα που δεν το έχουμε συζητήσει εδώ. Δηλαδή, να δούμε κατά πόσον η άμεση ενίσχυση είναι ενίσχυση εισοδηματική, ενίσχυση του εισοδήματο των αγροτών ή ε, σε ό,τι αφορά τον τζίρο, τον κύκλο εργασιών, γιατί δεν είναι το ίδιο και νομίζω ότι θα, είναι, θα πρέπει να είναι σαφής η συζήτηση. Έσοδα, εισόδημα, κύκλος εργασιών Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και αν περιορίζουμε το επίπεδο, το περιορίζουμε γιατί είναι στήριξη του εισοδήματο και όχι του κύκλου εργασιών. Αλλιώς θα μπορούσαμε επαόριστο να τα να στηρίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μπλοκάρισμα και πάβει να χρηματο, πάβουν να χρηματοδοτούνται οι μη ενεργοί ε, χτινοτρόφοι. Ε, η βασίλισσα της Αγγλίας, ο πρίγκιπας του Μονακό δεν παίρνουν χρηματοδότηση. Ε, λοιπόν, πρέπει να είναι σαφές. Δεύτερος στόχος, να έχουμε μια βιώσιμη, να μην πω πράσινη, εκείνη η γεωργική πολιτική. Βιώσιμη λοιπόν, υποστηρίξιμη, άρα με πρακτικές που θα δίνουν το δυνατότητα στη γεωργία να συνεχίσει με ε, και να επιτρέπει επίσης στη γεωργία να προσαρμοστεί στην αλλαγή του κλίματος. Και αυτή η δεύτερη πτυχή είναι καινούργια πτυχή. Το να μπει στον πρώτο πυλώνα νομίζω σημαίνει αλληλεγγύη μεταξύ Ευρωπαίων. Όλες οι χώρες δεν είναι ίσες απέναντι στα οικονομικά προβλήματα σε σχέση με τον προπολογισμό της χώρας τους. Σήμερα η Ελλάδα, η Ιρλανδία δεν έχουν τα ίδια μέσα για να στηρίξουν τους αγρότες τους σε σχέση με, τη Γεωργία, με την ε, Γερμανία και τη Γαλλία. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια συνέπεια, μια συνεκτικότητα και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε από κοινό αυτό το σχέδιο. Ο Μάρκ Ταραμπελά τώρα έχει το λόγο και μετά η κυρία Μαγκίνες. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να σας πω μια ιταλική φράση, μια φράση του Γκράμση που λέει όποιος δεν ξέρει που παίχνει, δεν ξέρει και που πάει. Θέλω να χαιρετήσω την δουλειά του Άλμπερτ Ντές που φυσικά δούλεψε για την έκθεση αυτή. Διαβάζοντα όμως την έκθεση ε, φοβήθηκα ε, διότι πρέπει να σας πω ότι κάποιο καιρό τώρα δουλεύουμε με βάση τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας που μας δίνει το δικαίωμα της συναπόφασης. Δουλέψαμε λοιπόν ε, στο πλαίσιο διαφόρων εκθέσεων με σημαντικά νοήματα, George Lyon, έκθεση George Lyon κτλ. Δεν λέω, προσπάθησε ε, ο Άλμπερντες, προσπάθησε αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα, όπως ανέφεραν στην άλφη 6, 10, 22, 25 παράγραφοι, η υποσημείωση για το σημείο 27 ή το σημείο 33 σε ό,τι αφορά τις μας παρεμβάσεις και τα λοιπά, αυτό το δίκτυο ασφαλείας. Ε, έχουμε κάποια προβλήματα με αυτή την ρευστότητα που θα συνεχιστεί βέβαια και στο μέλλον, αλλά μιλάμε για διασφαλίσεις αλλά για δημόσιες παρεμβάσεις γιατί περιορίζονται αυτό το δίκτυο ασφάλεια. Εγώ πραγματικά φοβάμαι, θα πρέπει να τροποποιηθεί η έκθεση. Εμεί θα συντάξουμε τροπολογίε και θα προσπαθήσουμε έτσι να δώσουμε με την έκθεση ένα συνεκτικό μήνυμα. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι με τι τροπολογίε τη έκθεση πρέπει να δώσουμε ω κοινοβούλιο ένα ισχυρό μήνυμα και δεν θα πρέπει το δικαίωμα συναπόφαση ε, ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο να καταπνιγεί ή να μετριαστεί. Διαβάζοντας εγώ ε, την έκθεση ήταν σαφής αυτά, σαφή αυτά που θέλει να πει, αλλά ε, από το σημείο 1 στο 58, ε, μία στις τρεις φράσεις μου δημιουργούν προβλήματα. δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Εγώ λέω, πρέπει το Κοινοβούλιο να δώσει ένα σαφές μήνυμα και αυτό θα είναι δύσκολο να το πετύχουμε νομίζω. Ευχαριστούμε κυρία Μαγκίνες και μετά κυρία Κασιμπερέσου. Ευχαριστώ, δεν έχουμε χρόνο πρόεδρε, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντές που ανέλαβε μια τόσο δύσκολη έκθεση αυτή που για όλους είναι το θέμα. Τόσο καιρό να ζητούμε μια σωστή κατεύθυνση και η έκθεση αυτή μας ανάγκασε να σκεφτούμε πιο προσεκτικά τι ακριβώς θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή την Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι σχεδόν ε, αδύνατο να επιτελέσει το έργο που ανέλαβε. Η μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτική φαίνεται ένα ανέφικτο ώστε να καλύπτουν τώρα τα ζητήματα που έχουμε τώρα επισημάνει συνάδελφοι σήμερα το απόγευμα. Δεδομένου δεν έχω πια χρόνο να κάνω κάνω την εξή παρατηρήσει. Δεν συμφωνώ συνήθω με τον κύριο Μποβέ, όμω τον ευχαριστώ για δύο αναφορέ του. Πρώτον, το ζήτημα τη βιώσιμη γεωργία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία. Αυτό είναι ένα ε, στόχο και θα πρέπει να τον επιδιώξουμε με μια ανάλογη μεταρρύθμιση τη πολιτική. Το δεύτερο σχόλιο του για την Ιρλανδία το σημειώνουμε με τα χαρά. Όμω υπάρχουν και άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να είναι σε κατάλληλη θέση να χρηματοδοτούν του γεωργού. Όμω να είμαστε ειλικρινεί. Νομίζω η Επιτροπή μα ανέκαθεν υπήρξε ειλικρινή. Όταν μιλάμε για κοινή γεωργική πολιτική, συζητούμε για 100% χρηματοδότηση με απευθεία πληρωμέ. Οπότε, οπότε αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε συμφωνήσει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε κάθε μα κίνηση να μην προκαλούμε στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά, ιδίω στην κοινή γεωργική πολιτική. Εκτιμώ λοιπόν ιδιαίτερα τα σχετικά σα σχόλια, κύριε Μποβέ. Εδώ λοιπόν αυτό που πρέπει να ορίσουμε είναι το greening, το πρασίνισμα λίγο καλύτερα. Το συζητούμε και δεν είμαι βέβαιο ότι σίγουρα το καταλαβαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Τέλο, θα πρέπει να σκεφτούμε του ορισμού τη ενεργή γεωργία. Εδώ πρέπει να δούμε τι συμβαίνει ακριβώ. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ μικροί γεωργοί που είναι ενεργοί, αλλά έχουν και άλλε ασχολίε από, από τι γεωργικέ του δραστηριότητε. Να το ξαναδούμε λοιπόν αυτό με μεγαλύτερη προσοχή και λεπτομέρεια. Και βεβαίω χρειαζόμαστε ένα μήνυμα συνεπέ και συνεκτικό. Αυτό θα προκύψει από τι τροπολογίε νομίζω που θα υποβάλουμε. Και θα φροντίσω και εγώ ίδια να αποβάλω τέτοιε. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι το εξή. Οι αρμόδιε αρχέ των 100 μελών είναι σαφώ οι πλέον υπεύθυνε και αρμόδιε για να αποφασίσουν για την υλοποίηση. Άρα χρειάζεται η διελεξία. Χρειάζεται έστω και εντό τη κοινά συμπεφωνημένη δομή με ό,τι μορφέ και αν προβλέψουμε. Αυτό το λέω στον ε, Άλμπερτ, Ευχαριστώ τον ξανά για την εντελεχή του έκθεση. Θα τη μελετήσουμε προσεκτικά και θα κάνουμε και τροπολογίε αναλόγω. Ευχαριστούμε, Μαρέιντ. Και τώρα η κυρία Γκαρσία Περέσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Νομίζω ότι συμφωνούμε στα βασικά όλοι οι σύντροφοι της Επιτροπής μας για τα γενικά ζητήματα, δηλαδή η εστίαση, συμπλήρωση στρατηγικής 2020, ανάγκη επαρκούς προπολογισμού, ανάγκη μέσων της αγοράς, ο ορισμός του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Ωστόσο, όπως και άλλους συντρόφους, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι στο πλαίσιο των προθέσεων ή των στόχων της απλούστευσης και της πρακτικής εφαρμογής των στόχων που θέτουμε, υπάρχει εντύπωση ότι ο αντίθετος στόχος εκπληρώνεται, δηλαδή αυξάνονται οι αμφιβολίες. Και σας αναφέρω ως παράδειγμα αυτό που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, σε σχέση με το άθρο 22. Αν μιλάμε για δύο πυλώνες πολύ καλά καθορισμένους, δεν καταλαβαίνω γιατί στη συνέχεια πρέπει να θέσουμε αυτούς τους όρους, μεταφορά, ε, συμπληρώματα κάποιων όρων σε, σε, από τον ένα πυλώνα στον άλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι λίγο ασαφές, είναι λίγο σκοτεινό. Και υπάρχουν και άλλα θέματα, φαντάζομαι όμως ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Πάντως, για άλλα, νομίζω ότι χρειάζεται και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση της Επιτροπής μας και να έχουμε έτσι και μια σταθερή θέση στο πλαίσιο και των προσεχών διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σημαντικότατο έργο που έχει επιτελέσει. Νομίζω η εκθεσή του επιβεβαιώνει κάποιες βασικές αρχές και είναι και κάποια άλλα θέματα για τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί το Ευρωκοινοβούλιο, όπω να αποβάλουμε κανόνες κοινού, ε, επαναλαμβάνοντα βέβαια την άποψη ότι δεν χρειάζεται επανακρατικοποίηση των πολιτικών, να υπερασπίσουμε τι ιστορικέ ανάγκε, την διοικητική απλούστευση, και μια αναθεώρηση που θεωρείται θεμελιώδου σημασία για την οικολογική συμμόρφωση εδώ, για του οικολογικού όρου. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με μια προσέγγιση ρεαλιστική, ακολουθωντα μια οικονομική, κοινωνική και ζωοτεχνική στάση ορθή. Εδώ λοιπόν το θέμα του εισοδήματο των γεωργών, της λειτουργίας της ε, αλυσίδας τροφή και το πώ καλύπτονται οι ανάγκε των καταναλωτών, όλα αυτά είναι σημαντική σημασία και πρέπει να καλυφθούν στην έκθεση. Πολλά είναι αυτά που να συζητηθούν, ιδίω του πρασινίσματος, του greening, της ε, οικολογικοποίησης. Αυτό το έχουμε συζητήσει λοιπόν ε, και με πολλούς ενδιαφερόμενους και είναι και κάτι που απασχολεί όλους μας τους πολίτες. Ε, για το θέμα αυτό ανακάλυψα ότι στη Γερμανία λόγου χάρη το θέμα αυτό φαίνεται να καλύπτεται από τον δεύτερο πυλώνα. Το ανακάλυψα μιλώντα με ενώσει ε, γεωργών. Ενώ στη Γαλλία θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορεί να βρίσκονται παρά στον πρώτο πυλώνα. Και αυτό επειδή μπορεί να υπάρχουν χρήματα που αποδίδονται στο δεύτερο, αλλά ε, πρέπει κάτι να γίνει και στον πρώτο. Εδώ λοιπόν τα πράγματα φαίνονται αρκετά μπερδεμένα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι σκέφτονται οι διάφορε κοινέ μα γνώμε στι διαφορετικέ χώρε για να δούμε πώ θα επιλύσουμε κάποια θέματα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ολοκληρώνουμε με τον ίδιο τρόπο την οικολογικοποίηση αυτή. Όπω ε, επίση την επιστηστική ασφάλεια, βλέποντα πώς ε, έχουν συνταχθεί κάποια εδάφια, νόμιζα ότι είχαμε συνεννοηθεί. Τελικά δεν εννοούμε φαίνεται τα ίδια πράγματα πάντοτε. Γι' αυτό λοιπόν, Πρόεδρε, θα πρέπει να φροντίσουμε να υποβάλουμε τι τροπολογίε, αφού όμω προηγουμένω συζητήσουμε μεταξύ μα την Επιτροπή, διευκρινίσουμε κάποια πράγματα και ε, εξακριβώσουμε τι εννοούμε μεν και ιδέ με συγκεκριμένου όρου. Διότι την ώρα των τροπολογιών θα ανακαλύψουμε που έχουν γίνει ανασυνεννοησίε και ότι δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα μιλώντα με τι ίδιε λέξει. Ευχαριστούμε. Μισελ, ο κύριος Γιάρ. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή. Βεβαίως η έκθεση αυτή δεν είναι απλή και το έργο που ανέλαβε είναι μεγάλο. Δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, δεν θα πρέπει να αγνοούμε τα στοιχεία στα οποία συμφωνούμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα των πράσινων μέτρων, το greening και να βρούμε και τα αναγκαία, τις αναγκαίες πιστώσεις. Όμως πρέπει να είμαστε και σαφείς στους στόχους μας. Καταρχάς πρέπει να, είναι, να μην είναι γραφειοκρατικά τα μέτρα αυτά και ε, δεν νομίζω ότι ε, τα μέτρα αυτά έχουν την ίδια τιμή, την ίδια αξία σε όλα τα κράτη. Σε ορισμένα μπορεί να είναι 15 ευρώ ένα στοιχείο και σε άλλο να είναι 25 ευρώ. Επίσης ε, δεν πρέπει αυτά τα πράσινα μέτρα, αυτή η πράσινη πτυχή να διακυβεύσουν ε, άλλα περιβαλλοντικά μέτρα τα οποία οι παραγωγοί εφαρμόζουν θελούσια, προαιρετικά. Και θα πρέπει επίσης και να προσέξουμε ε, πώς τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Αυτά λοιπόν, αυτό λοιπόν το πρασίνισμα γενικά πρέπει πιστεύω να μπει στο δεύτερο πυλώνα, στη δεύτερη στήλη. Δεν είναι υποχρεωτικό να μπουν στην πρώτη στήλη Λοιπόν, να σκεφτούμε τι στόχους θέλουμε να επιτύχουμε με την πράσινη πτυχή και τι θέλουμε η παραγωγή να κάνουν προς αυτό το σκοπό. Επίσης, η πολιτική δεν μπορεί να εκφράζει επιθυμίες. Ε, πρέπει να ε, εφαρμόσουμε μέτρα βιώσιμα και όχι ιδεατά. Ευχαριστώ στο Στρασβούργο. Θα έχουμε περίπου μία-μία μισή ώρα χρόνο για να ε, συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Ε, ξέρετε ότι 14 Μαρτίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και πρέπει να υποστηρίξουμε τον Άλμπερτ και σαφώς χρειάζεται μία συζήτηση στην εβδομάδα του Στρασβούργου. Ευχαριστώ και εγώ τον Άλμπερτ για το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Δεν πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εγώ πιστεύω ότι η επισητιστική επάρχεια, βιοπικιλότητα και κλιματικές αλλαγές είναι οι απόλυτες προτεραιότητες. Είχα μία ολόκληρη δέσμη ερωτήσεων, αλλά λόγω της έλλειψης χρόνου θα συγκεντρώσω την προσοχή μου σε μία-δυο ερωτήσεις. Λέει στα εκτιμώντας ότι οι γενικοί στόχοι της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν πρέπει να υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών. Το ερώτημά μου, οι άμεσες πληρωμές έχουν ως στόχο να δίνουν τη δυνατότητα ενός συγκεκριμένου εισοδήματος στον παραγωγό. Εάν τώρα αλλάξουμε τη διαμόρφωση της πρώτης στήλη, διακυβεύουμε αυτό το στόχο. Και κάτι άλλο ακόμα. Ε, πιστεύω ότι τα, τα, τα, οι πιστώσεις οι οποίες ήταν διαθέσιμες για τα εισοδήματα των, των παραγωγών μπορούν να εξαφανιστούν με μονοκονδυλιά. Γι' αυτό παρακαλώ προσέξτε πάρα πολύ τα προτινόμενα μέτρα. Επίσης δεν θα πρέπει να δημιουργήσει μεταρρύθμιση το νέο καθεστώς παραγωγούς πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ε, πολλές φορές υπόθηκε ότι πολλές φορές η συγχρηματοδότηση δεν είναι δυνατή. Ε, αφού θέλουμε μια κοινή γεωργική πολιτική, γιατί δεν μπορούμε να επιτύχουμε και κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Επίσης θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος στην παράγραφο 36 τι εννοούμε με, μέτρα στρέβλωσης των αγορών. Ευχαριστώ. Δευτέρα στις 7 Μαρτίου η συνεδρίασή μας μπορεί να γίνει στις 7 το βράδυ την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Μαρτίου. 7 το βράδυ, μία-μία μισή ώρα για συζήτηση. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι... Θα, θα ήθελα να εκφράσω τις απόψεις μου και δεν καταλαβαίνω γιατί υποχρεώνω που με πιέζεται για ένα λεπτό αφού ακούσαμε τόσους προλαλήσανες να μιλάνε εν Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να συμφιλιώσουμε όλες τις διαφορετικές μας απόψεις ε, σε μια ολοκληρωμένη έκθεση με τόσες διαφορές που υπάρχουν βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά. Η πολιτική της ε, Λετωνίας βασίζεται στο στοιχείο της δικαιοσύνης, του δίκαιου, του θεμητού. Πρέπει όλα τα μέτρα που αποφασίζονται να είναι δίκαια προς όλους τους παραγωγούς. Και ε, γι' αυτό χαιρετίζω την πρόταση να ορίσουμε τα μέτρα αυτά στο κατώτερο επίπεδο αναεκτάριο. Επίσης, ε, το ιδέα του capping των πληρωμών αναεκτάριων πιστεύω ότι είναι επίσης σωστή το ανώτατο όριο πρέπει να είναι 75% του μέσου όρου πληρωμών στην Ευρώπη. Επίσης η μεταβατική περίοδος πιστεύουμε δεν πρέπει να είναι πέραν των τεσσάρων ετών. Και στην προηγούμενη μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής, της κοινής πολιτικής είχαμε μία τετραετή μεταβατική περίοδο. Η Λετωνία ε, θέλει να εφαρμοστούν ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια στην διάθεση των πιστώσεων. Καταρχάς το ε, ΑΕΠ το εθνικό ΑΕΠ ή ε, το ποσό, οι δαπάνες που χρειάζονται για τη λειτουργία μιας ε, μονάδας, μιας εκμετάλλευσης να εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια έτσι ώστε παρόλο που υπάρχουν διαφορές να μπορέσουμε να τις γεφυρώσουμε. Κάνε... Κοιτάξτε, έχουμε χρόνο και τη Δευτέρα ποιος θα θέλει να μιλήσει τώρα μπορεί να το κάνει τη Δευτέρα. Ähm, θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη ότι είχαμε μία οικονομική κρίση στην Ευρώπη μεγάλη. Αυτή τη στιγμή ε, έχουμε επίσης και μεγάλα πολιτικά γεγονότα εκτός Ευρώπης τα οποία θα έχουν επιπτώσεις στη γεωργία διότι ο γεωργικός τομέας είναι παγκόσμιος και συνέχεια αναφερόμαστε στο τι προσδοκίες, τι θέλουμε, τι πρέπει να ε, ε, παρουσιάσουν οι παραγωγοί. Όμως στόχος μας πρέπει να είναι η οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και δεν θα πρέπει να εκφράζουμε υπερβολικά πολλές επιθυμίες και προσδοκίες, αλλά να είναι ρεαλιστικές. Ο κύριος Καλινός και μετά ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι εξαιρετική η έκθεση του κυρίου Ντέ. Απαντά σε πολλά ζητήματα, αλλά υπάρχει και μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, η οποία είναι μέγιστη σημασία και μόνο εν μέρη ε, απαντάται. Είναι δηλαδή ανταγωνιστικότητα τη γεωργία στην Ευρώπη. Υπάρχει εδώ διεθνή ανταγωνισμό. Και αυτό πρόσφατα φαίνεται να μα δυσκολεύει ιδιαίτερα εισαγωγέ από τρίτε χώρε θα έπρεπε να γίνονται με κριτήριο το αν έχουν ε, ισότιμες προδιαγραφές για τη ζωική ζωή όπως η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν οι προδιαγραφές αυτές να πληρούνται, όχι μόνο να τις αναφέρουμε, ούτε μόνο να συζητούμε τι επιδοτήσεις θα δίνονται στη γεωργία. Πρέπει να έχουμε αντικειμενικά κριτήρια εδώ πέρα. Εδώ υπάρχουν κάποιες ε, περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε τι διαφωνίε. Είναι διαφορετικέ οι γεωργικέ συνήθειε σε πολλέ χώρε. Όμω πρέπει γι' αυτό ακριβώ το λόγο να εξεύρουμε αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό λοιπόν που. Ε, μας απασχολεί είναι ακριβώς σε τέτοια κριτήρια να βασιστούμε για τις άμεσες πληρωμές. Ευχαριστούμε ο κύριος Σμιτ και μετά Κέστιγκερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομε παρατηρήσεις. Δεν θα επαναλάβω όσα ήδη υπόθηκαν για την ανάπτυξη της υπαίθρου ε, και τις λιγότερο ευνοούμενες περιοχές. Εδώ ανησυχούμε κάπως για τον κατάλογο των δεσμευτικών μέτρων που θα αντικαταστήσουν προηγούμενες ε, δράσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θέλουμε να υποθεί σαφώς ότι το καλύτερο, το πλέον καινοτόμο είναι να εγκρίνονται πρόγραμμα, προγράμματα που επιτρέπουν τη μέγιστη ευελιξία και την επιλογή από τοπικού φορεί. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να είμαστε σαφεί ε, στο πώ θα προωθηθεί αυτό το μέτρο και για τα προγράμματα υπέρ των ε, λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Αυτό για τι ευάλωτε περιοχέ είναι ιδιαίτερε σημαντικό πρέπει ανάγκη ανάγκε των μικρότερων γεωργών να ληφθούν υπόψη σε όλη αυτή η μεταρρύθμιση και τι προτάσει μα την κοινή γεωργική πολιτική. Θα φροντίσουμε λοιπόν να υποβάλουμε τροπολογίε ώστε και το στοιχείο αυτό να τονιστεί επαρκώ στην έκθεση και να προωθηθεί. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σμιτ, ήσασταν τέλειο στο χρόνο ομιλία. Στο χρόνο Ο κύριος, η κυρία Γκέτιγκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το συζητάμε σήμερα για το greening στην πρώτη στήλη να μην επιδεινωθεί η θέση χωρών που ήδη έχουν προσφέρει πολλά στο γεωργικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε όταν συζητάμε για τον πρώτο πυλώνα ότι πολλές χώρες ήδη έχουν συμμορφωθεί με την πολλοπλή, σέβονται την πολλαπλή συμμόρφωση και έχουν εφαρμόσει πολύ επιτυχώς ε, μέτρα του γεωργικού τομέα. Αυτό το οποίο πιστεύω πρέπει να προσέξουμε είναι ο τομέας της διαχείρισης κινδύνων, του ρίσκου και βλέπουμε τι συμβαίνει στις γεωργικές αγορές ε, σήμερα και βλέπουμε τις υψηλές ε, τιμές ε, που υπάρχουν στις αγορές ζωοτροφών και τι επιπτώσεις έχουν ιδίω στη χειροτροφία. Ε, έχουμε, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τους κερδοσκόπους και πρέπει να εμποδίσουμε τη κερδοσκοπία με κάθε μέσο. Ε, καλωσορίζω τα μέτρα τα οποία ενισχύουν τις μειονεκτικές περιοχές και τις ορεινές περιοχές και επίσης υποστηρίζω τα πριμ για ε, τις θυλάζουσες αγελάδες και τονίζω ότι ε, και ο τομέας των νέων παραγωγών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής δεν είμαι σίγουρη ότι τα μέτρα που προτείνει στη δεύτερη στήλη επαρκούν ε, ιδίω για τους νέους γεωργούς. Μήπως θα πρέπει να εφαρμόσουμε πιο θαραλέα μέτρα για αυτούς. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπλόσεβιτς και ο κύριος Άγνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντες, όπως και άλλους, διότι η έκθεση αυτή αποτελεί μια βάση, ένα θεμέλιο σταθερό για, τα, για τη συνέχεια του έργου μας. Νομίζω ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και φαίνεται εδώ να δίνει την απαραίτητη μέρημνα στο, στο να εξασφαλίσει ένα μέλλον για τη γεωργία στην Ευρώπη. Το θέμα είναι όμως πώς θα εξαλείψουμε τις μεγάλες ανισότητες μεταξύ παλαιών και κρατών μελών, ιδίως στον τομέα των απευθείας πληρωμών. Δεν είναι σαφές ποιο θα είναι, ποια θα είναι η, μορφή, μελλοντική μορφή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει πολλά στοιχεία να καλυφθούν από την πολιτική αυτή, αλλά οι διαφορές των χωρών δεν μπορεί παρά να οφείλονται και σε διαφορετικές γεωργικές συνήθειες. Και φυσικά υπάρχουν επιπτώσει στι άμεσε πληρωμέ και στο επίπεδο τη στήριξη. Αυτό όμω το επίπεδο τη στήριξη δεν πρέπει να βασίζεται στο, στη χώρα προέλευση των Γεωργών. Επίση πρέπει να προβλεφθούν πόροι ίσοι για όλου του Γεωργού. Έχουμε δει ανισότητα στην κατανομή των πόρων. Κάποιες χώρες είναι θύματα αρνητικής μεταχείρισης σε σχέση με άλλες και διακριτικής μεταχείρισης. Σε κάποιε χώρε υπάρχουν γεωργοί που ακριβώ λόγω αυτή τη διακριτική μεταχείριση πήραν λιγότερα ποσά. Εάν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει ισότητα και δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Στην, κοινή, στη νέα κοινή γεωργική πολιτική, λοιπόν, θα πρέπει να αναπτύξουμε πραγματικά κοινά κριτήρια για τη στήριξη των γεωργών, γιατί δεν θέλουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Ο κύριο Άγνιου. Άλμπερτ, μ' Εκτός μικροφώνου κύριο Άγνιου, οπότε δεν ακούγεται. Albert, Άγνιο, από τα μέλη σου κατάλαβα ότι έχεις γίνει σοσιαλιστής. Ακόμη και ο Βρετανό Υπουργό Γεωργία ε, ανέφερε ω σοσιαλιστή την Πέμπτη. Μπορεί να το επιβεβαιώσει, να το ε, διαψεύσει, αλλά το θέμα είναι και η πηγή από την οποία προέρχεται το σχόλιο. Τέλο πάντων, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα την, για την έκθεση αυτή. Εσύ όμω είσαι ο πρώτο από του βουλευτέ, θα πρέπει εδώ να με υποστηρίξει στη, στα σχόλια που κάνω και εγώ για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι ε, σαφέ ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αύξηση τη θερμοκρασία του πλανήτη και ελπίζω να με στηρίξει μελλοντικά στο θέμα αυτό. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να συμφωνήσουν στην συγχρηματοδότηση του δευτέρου πυλώνα. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει πολύ λίγα ποσά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Οπότε στο μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι τέτοιο, ιδίω για του Βρετανού προλογουμένου που τόσο πολύ έχουν επιβαρυνθεί. Δεν μπορούν να δεχτούν να μπει και άλλο χέρι στην τσέπη του και να του πάρει χρήματα για τη συγχρηματοδότηση του δεύτερου πυλώνα. Ε, τώρα, για το κάπινγκ. 59 δευτερόλεπτα, Πρόεδρε. Ε, Όπω είδατε, σεβάστηκα το χρόνο μου. Ευχαριστούμε, κυρία Άγνιο. Κύριο και κυρίες και μετά, κλάσ. Moje Ευχαριστώ. Ο δεύτερος ε, πυλώνας ε, στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν βλέπω όμως πώς θα συμπληρώνει τον πρώτο πυλώνα, την πρώτη στήλη στον τομέα του εξυγχρονισμού. Χρειαζόμαστε επιγόντως μέτρα εξυγχρονισμού. Στο παρελθόν οι ανισότητες του, της, του, πρώτης στήλης εξομαλύνονταν με μεταφορές από τη δεύτερη στήλη ιδίω για τις νέες καινούργιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί φοβόμαστε τις επεμβάσεις στις γεωργικές αγορές. Εάν δεν παρέμβουμε ε, θα αποτύχουμε, ε, όπου χρειάζεται δηλαδή μια παρέμβαση. Εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν θέλει να κάνει μια μεταρρύθμιση μόνο στα χαρτιά. Ουσιαστικά δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ τον Άλμπερτ που πρέπει να συγκεράσει όλα αυτά τα θέματα και χαίρομαι που προχωράμε στη συζήτηση βήμα προς βήμα. Ε, τα κράτη-μέλη συνήθως εμένουν στη στάση τους, ε, δεν δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο λιγμών λένε πάντοτε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα, τις απαραίτητες πιστώσεις ε, και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ισχυρή πρώτη στήλη. Ο Άλμπερ Ντες δικαιολογεί όλα του τα επιχειρήματα σαφέστατα, λέει ότι χρειαζόμαστε περιφερειακά μέτρα τα οποία θα πρέπει να προσαρμόζονται βεβαίως ε, αντίστοιχα σε κάθε περιφέρεια ε, στο θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικά, διαφορετικές αντιμετωπίσεις από τα κράτη-μέλη. Ε, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις ε, της κοινή διορικής πολιτικής ε, για την υγιή ανάπτυξη του γεωρικού μας τομέα και για να εξασφαλίσουμε τις επαρκείς πιστώσεις. Ευχαριστούμε κυρία Κλάς. Ο κύριος Βότσιεβός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο προλαλή σα μίλησε για ισότητα, αδελφότητα και τα λοιπά. Και είπε δεν έχουμε ισότητα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Έχουμε ισότητα και μάλιστα έχουμε δύο ισότητες. Έχουμε μία ισότητα για κάποιους, τα κράτη-μέλη συγκεκριμένα, και μια άλλη ισότητα μια νέα προσέγγιση δηλαδή, μια άλλη προσέγγιση για τα νέα κράτη-μέλη. Μιλάμε για την Ευρώπη των ε, δύο ταχυτήτων, αλλά έχουμε και την Ευρώπη των δύο ισοτήτων. Τουλάχιστον στην κοινή γεωργική πολιτική. Τώρα, ό,τι και να κάνουμε με τη μεταρρύθμιση, θα πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή την Ευρώπη των δύο ισοτήτων. Θα πρέπει να πετύχουμε μια ενιαία Ευρώπη, όπου όλοι οι πολίτε και όλες οι χώρες αντιμετωπίζονται ισότιμα. Φυσικά και θα πρέπει να υπάρξουν διαφορές άμεση πληρωμές για διαφορετικούς λόγους. Αλλά όχι λόγω της χώρας στην οποία καλλιεργεί ο κάθε αγρότης. Πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις διαφορές αυτές να τις υπερκεράσουμε γιατί ήταν άδικες είναι άδικες. Μιλάμε για ίσες πληρωμές και δίκαιες πληρωμές. Κατανομή των πόρων, των κονδυλίων, πρέπει να είναι δίκαιη. Αλλά πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση για να υπάρξουν οι δίκαιες αυτές πληρωμές, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ποτέ δεν θα έχουμε δικαιοσύνη. Παραλαμβάνω λοιπόν, θέλω όλοι να έχουμε ισότιμη μεταχείριση για να μπορέσουμε να έχουμε μια δίκαιη πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από όλου γιατί χρειάστηκε να τρέξουμε τόσο πολύ. Αλλά αν συμφωνεί ο Άλμπερτ, και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και από του εκπροσώπου τη Επιτροπή, είχαμε τέσσερι διευθυντέ σήμερα μαζί μα. Σκεφτήκαμε να γίνει το εξή, Άλμπερτ. Θα ξαναβρεθούμε στο Στρασβούργο τη Δευτέρα στις 7. Στις 7 το απόγευμα και εκεί θα δώσουμε απευθείας το λόγο στον Άλμπερτ ώστε να ανταποκριθεί σε όλα τα σχόλια που έγιναν σήμερα. Εκεί το λόγο θα έχουν και εκπρόσωποι της Επιτροπής που με την συγκεκριμένη ευκαιρία και με λίγο περισσότερη ηρεμία θα μπορούν να μας πούν την άποψή τους τα λίγα λεπτά που μας έμειναν να τα αφιερώσουμε πάρα πολύ γρήγορα στα όσα έχουμε να πούμε συντονιστές. Άλμπερτ, σε σένα ο λόγος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα, το μόνο που έχω να πω είναι να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν το λόγο δεν με πειράζει καθόλου όταν ακούγονται αυστηρές ε, κριτικές εκ μέρους των συναδέλφων. Έχω διαπιστώσει πολλές φορές ε, ότι ο όρος δίκαιο, δικαιοσύνη ε, σηκώνει πολλαπλές ερμηνείες. Το έχω διαπιστώσει αυτό στις περισσότερες συζητήσεις που έχω κάνει μέχρι τώρα έχω διαπιστώσει αποκλίνουσες απόψεις. Σας συστήνω να διαβάσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδος όπου θα διαπιστώσετε πόσο αποκλίνουν οι απόψεις. Εγώ θα προσπαθήσω να συγκεράσω τις ε, παρατηρήσεις και τις απόψεις ε, που άκουσα για να μπορέσω να, να τις ενσωματώσω επικοδομητικά στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ Άλμπερτ, ευχαριστώ όλου, ευχαριστώ και του εκπροσώπους τη Επιτροπή. Θα βρεθούμε στο Στρασβούργο για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Και τώρα σα παρακαλώ, οι συντονιστέ, ένα μόνο λεπτό για να αποφασίσουμε το πρώτο σημείο.